Καλημέρα σας. Θα μιλήσω ισπανικά. Παρακαλώ βάλτε τα ακουστικά σας. Αρχίζουμε λοιπόν τη σημερινή συνεδρίαση με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν έχετε παρατηρήσεις, εγκρίνεται. Ανακοινώσεις από την Προεδρία δεν έχουμε, οπότε και θα περάσουμε αμέσως στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι μια δημόσια ακρόαση κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράση, επιλογέ πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε περίπτωση ανάκληση τη επικύρωση εκ μέρου των Ηνωμένων Πολιτειών τη Αμερική. Αυτή τη συμφωνία τη γνωρίζουμε κοινώ ω πυρηνική συμφωνία με το Ιράν, αν και ονομάζεται κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράση. Είναι σημαντικέ οι επιπτώσει για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε περίπτωση που αποσυρθούν οι Ηνωμένε Πολιτείε και επιβάλλουν κυρώσει. Θέλω ε, να ε, καλωσορίσω τον κύριο Αντεμπαχάρα από το Κάνε και Europe και την κυρία Γκέραν Μάγε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων. Στις 16 Φεβρουαρίου 2018 ο πρόεδρος Τραμπ παρουσίασε το Κογκρέσο και στους συμμάχους μία ε, πρόταση ε, που πρέπει να εγκριθεί μέχρι τις 12 Πέμπτου του 2018. απειλεί να επανέλθουν οι κυρώσεις στο Ιράν εάν δεν είναι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα το διαπραγματεύσεων. Στις τελευταίες εβδομάδες ε, έδωσε και ανησυχητικά σημεία με κάποιους διορισμούς που έκανε ο κύριος Τραμπ ε, και είναι ανισχυτική για το μέλλον της συμφωνίας με το Ιράν. Το Κοινοβούλιο μας επανειλημμένα έχει τονίσει την απόλυτη και πλήρη στήριξή του προς την συμφωνία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν διαφωνούμε με το Ιράν ή ότι εγκρίνουμε την εσωτερική κατάσταση στη χώρα, την πυραυλική, πολιτική κλπ. Αλλά θεωρούμε αυτά τα σημεία διαφωνίας ότι πρέπει να είναι εκτός της συμφωνίας και ο κόσμος δεν πρόκειται να είναι πιο ασφαλής αν δεν υπάρχει συμφωνία, μάλλον το αντίθετο. Η εισαγωγή κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξει απολύτως ε, ευρωπαϊκές εταιρείες που έχουν επενδύσει στο Ιράν. Δεν θα πλήξει ε, άμεσα τις ε, εξαγωγές πετρελαίου από το Ιράν. Τι θα μπορέσει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να προστατεύσει τις ευρωπαϊκές εταιρείες που έχουν επενδύσει στη χώρα. Τι θα γίνει με την οικονομία του Ιράν. Ο πρόεδρος Ροχανή, ε, αφού του ανέλαβε, έχει συσφίξει τις σχέσεις με την Κίνα, την Ινδία, το Πακιστάν, οικονομικές και εμπορικές και το Αζερβαϊτσα. Αυτό άρχισε ήδη από την εποχή των διεθνών κυρώσεων. Τώρα, ποιες θα ήταν οι γεωπολιτικές και οι γεωοικονομικές επιπτώσεις της επαναφοράς των κυρώσεων. Θα δούμε να γραμμίζεται ακόμα περισσότερο με την Κίνα και με τη Ρωσία. Αν αποσυρθούν ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε από τη συμφωνία, τι θα γίνει. Ορισμένοι λέγουν ότι η κυβέρνηση Ρόχανη ε, θα σταματήσει να εφαρμόζει το πρωτόκολλο της μη διάδοσης, ενδίδοντας στα γεράκια και ε, προχωρώντας σε όξυνση. Τυπικά μεν θα τηρούσε τη συμφωνία και δεν θα μπορούσαν οι υπόλοιπες ε, χώρες ε, με τη συμφωνία να φέρουν κυρώσεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας είπε ότι το Ιράν θα απαντήσει με σοβαρό και αναλογικό τρόπο σε περίπτωση που επαναφέρουν τις κυρώσεις στις Ηνωμένες Ορισμένοι πυρογνώμονες λέγουν ότι το Ιράν θα μπορούσε να επιλέξει αυτή ακριβώς επιλεκτική ε, μη εφαρμογή ε, της συνθήκης μη διάσωσης. Αυτό το σενάριο είναι πιθανό. Ποια θα ήταν η πιθανή λοιπόν ε, ιρανική αντίδραση σε περίπτωση που αποσυρθούν οι ΥΠΑ από τη συμφωνία. Τι θα γίνει με τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων γενικότερα. Απαντήστε σας παρακαλώ σε αυτή την ερώτηση σε άλλες που θεωρείτε σκόπιμες για να καταλάβουμε καλύτερα πώς θα απαντήσουμε σε αυτή την όξυνση, την πιθανή. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Αντεμπαχά ε, για μια πρώτη παρέμβαση 10 με 15 λεπτά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα μιλήσω αγγλικά. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Να ευχαριστήσω το προσωπικό της γραμματείας που διοργάνωσε την εκδήλωση αυτή και ευχαριστώ και τον συνάδελφο για την παρουσίαση. Το σημερινό μας θέμα είναι ιδιαίτερα επίκαιρο. Αυτό θα μπορούσε να πει κανεί για κάθε συζήτηση με το Ιράν την τελευταία πενταετία. Γιατί διότι διαρκώς βρίσκεται στην επικαιρότητα η συζήτηση της ευρωπαϊκής θέσης ε, σε σχέση με το Ιράν. Όταν μιλάμε για την άρση της πιστοποίησης όμως έχουμε καθυστερήσει. Η άρση της πιστοποίησης συνέβη τον Οκτώβριο. Πρέπει να πω, είναι καθαρά εσωτερικό θέμα των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ήδη ε, αρνηθεί να πιστοποιήσει τη συμμόρφωση του Ιράν. Και τώρα βλέπουμε ε, την η προθεσμία του 12η Μαΐου, όπως είπε ο πρόεδρος, ε, τότε που θα μπορούσε να επανεισάγει κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών ο πρόεδρος. Εγώ βρέθηκα στην Τεχεράνη και μίλησα με υπευθύνου χάραξη πολιτική εκεί και μπορώ να σα πω ότι δυσκολευτήκαμε να υπερασπίσουμε τι ευρωπαϊκέ θέσει. Ευχαριστώ να αναλύσω λίγο σε εσά ε, τι ευρωπαϊκέ ε, πιθανέ θέσει. Η Ελή και εγώ αποφασίσαμε να μοιραστούμε την παρουσίαση. Εγώ θα σας δώσω τα... μια γενικότερη εικόνα της κατάστασης των διακυβευμάτων ε, από ευρωπαϊκή άποψη και μετά θα, η συνάδελφός μου η Έλλη θα μπει σε, στις λεπτομέρειες για το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν θέλουμε απλά να σώσουμε ε, την JCPOA. Αν, πάμε, αν δούμε στο παρελθόν και δούμε τι μας έχει προσφέρει ε, όσον αφορά τη σημερινή κατάσταση, θα πρέπει να ανατρέξουμε στο 2003, στην αρχή αυτών των διαπραγματεύσεων. Ας θυμηθούμε ποια ήταν τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκτοτε. Και πιστεύω ότι έχουν τρεις διαστάσεις, ε, βάσει των οποίων θα κάνω και την παρουσίασή μου. Πρώτο συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η πρόληψη ε, κατασκευής μιας πυρηνικής βόμβας από το Ιράν. Το δεύτερο συμφέρον, όπως και το 2003, είναι το να προλάβουμε άλλο ε, αυτό ε, κάτι που μας ανησυχεί σήμερα, να διαβάσει κανείς αυτά που έγραψε στο Twitter ο Τραμπ. Και τρίτον, ε, θέλει να δείξει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι έχει κάποιο βάρος στο παγκόσμιο σκηνικό. Αυτό συνέβαινε το 2003 και συμβαίνει και σήμερα. Για το πρώτο σημείο λοιπόν, το πρώτο συμφέρον, το πρωταρχικό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προλάβει ε, την κατασκευή ε, πυρηνικής βόμβας από το Ιράν. Έχουμε ένα εργαλείο στην JCPOA που είναι ύψης της σημασίας. Δεν είναι απλά για να υπάρχει, αλλά και για να υλοποιείται αυστηρά. Η συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αλλάξει εστίαση. Αντί για την υλοποίηση της JCPOA ουσιαστικά εξετάζει την εκθέση της ΔΟΕ που ε, επικυρώνει όχι τη συμμόρφωση του Ιράν. Κατά κανέναν τρόπο όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να κάνει τα στραβαμάτια όσον αφορά τα συμβαίνουν στο Ιράν ώστε απλά να κολακεύει το Ιράν και να διατηρεί ε, μία ε, παρουσία αυτού του γράφου εργασία το οποίο χρειάζεται διαρκή ενημέρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξετάζει την υλοποίηση της JCTOA διαρκώς να πραγματοποιεί επιθεωρήσεις κάθε φορά που υπάρχει υποψία ότι πρέπει να γίνει επιθεωρήση κάποιες τοποθεσίας και τα παρεμφερεί. Το δεύτερο κομμάτι της ε, υλοποίησης της JCTOA ε, σχετίζεται με αυτό που ονομάζουμε sunset clauses. Ε, ξέρουμε ότι έχει χρονικό όριο η συμφωνία αυτή διαφορετικά δεν θα είχαμε μια κοινή συμφωνία εθελοντική από πλευρά του Ιράν ε, για περιορισμό του ε, πυρηνικών ε, μέσων ακόμη και αν υλοποιηθεί πλήρως η GCTOA για 10-15 χρόνια πρέπει να ξέρουμε ότι το Ιράν θα είναι διαφορετικό από την εποχή πριν τη συμφωνία. Πολλέ από τι συζητήσει που σχετίζονται με τι ρήτρε εκπνοή, αυτέ τι sunset clauses, είναι ότι το Ιράν στη συνέχεια θα είναι ελεύθερο να επιδιώξει ένα πυρηνικό πρόγραμμα σε βιομηχανική κλίμακα και θα μπορεί να φτιάξει ε, πυρηνική βόμβα. Αν όμω ε, έχει υλοποιηθεί η JCTOA θα έχει, το, θα έχει κυρώσει το αρχικό πρωτόκολλο το Ιράν και θα συνεχίζει να είναι ε, πλήρες μέλος της σύμβασης μη διάδοσης υπό το πλαίσιο αυτού ε, της διασφάλισης. Καλό είναι λοιπόν να ξεκινήσουμε μια συζήτηση και διατλαντικά περί του τι θα σημάνει ε, η εκπνοή της JCTO κάποια στιγμή στο μέλλον. Αυτός ο διαλόγος θα πρέπει να εστιαστεί όχι μόνο στο Ιράν, αλλά και στη, στη συγκεκριμένη περιφέρεια και τις διάφορες πλευρές που συμμετέχουν εκεί. Ε, το περιφερειακό περιβάλλον εκεί θα μπορούσε να περιλαμβάνει τομεί ε, ε, προτύπων που έχουν συμφωνηθεί από κοινού και που οδηγούν στη διαδικασία κύρωση του πρωτοκόλλου, του πρόσθετου πρωτοκόλλου στην περιοχή. Και αναφέρομαι ουσιαστικά στον Περσικό κόλπο. Να προσπαθήσουμε δηλαδή να βρούμε τρόπους δεσμευτικούς για τις τοπικές δυνάμεις σε θέματα μη διάδοσης με τρόπου που δεν υπήρχαν, ε, δεν υπήρχαν πριν το JCPOA. Πρώτη προτεραιότητα, όπω είπα, είναι να προλάβουμε την κατασκευή βόμβα. Όπω γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, αυτό δεν αφορά μόνο το Ιράν και η Σαουδική Αραβία επίση ε, έχει αναφέρει ότι υπάρχει ενδεχόμενο να αποκτήσει πυρηνικό όπλο σε περίπτωση που αποκτήσει τέτοιο το Ιράν. Ε, όσο το βρίσκεται υπό το GCTOA, η Σαουδική Αραβία δεν πρόκειται ποτέ να αγοράσει κάτι τέτοιο. Η, η Σαουδική Αραβία είναι μέλος ε, της ε, συμφωνίας μη διάδοση και πρόκειται να αγοράσει δούμε, ένα μη στρατιωτικό πυρηνικό πρόγραμμα ώστε να αποκτήσει δυνατότητε εμπλουτισμού. Στο πλαίσιο αυτό, ο περιφερειακό διάλογο είναι σημαντικό ώστε να αποφύγουμε την κατασκευή οποιασδήποτε πυρηνική βόμβα ε, στην ε, χώρο του Περσικού κόλπου. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει, ο διάλογο θα πρέπει να περιλαμβάνει και τη μη στρατιωτική πυρηνική ενέργεια. Αυτό είναι σημαντικό ώστε οποιοδήποτε σαουδικό πρόγραμμα να είναι βέβαιο ότι συνάδει με τη Συμφωνία Μη Διάδοσης και με τα ε, διασφαλίσεις και οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να συνεργαστούν με τους Αμερικανούς ώστε να δουν ε, ποια θα είναι η συμμετοχή των ε, Αμερικανικών εταιριών στην, στο Σαουδικό πρόγραμμα. Α θυμηθούμε την υποστήριξη στο Ιρανικό πρόγραμμα από του Αμερικανού και η συζήτηση αυτή για τι δυνατότητε εμπλουτισμού. Όλα αυτά είναι σημαντικά για να καταλάβουμε πώ έχουν τα πράγματα σήμερα στο αναδυόμενο ε, σαουδικό ε, πυρηνικό πρόγραμμα. Το τελευταίο σημείο ε, αφορά τον περιφερειακό διάλογο. Υπήρξε μια πρόταση από τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν στην τελευταία διάσκεψη ασφαλείας νωρίτερα φέτος ο οποίο αναφερόμένο στο ψήφισμα 598 των ε, Ηνωμένων Εθνών για το τέλος του πολέμου Ιράκ-Ιράν ε, ε, αναφέρθηκε στη, ότι πρέπει να γίνει ένα διάλογο Το άλλο σημείο που είπα που αφορά την αποφυγή του πολέμου είναι κατεπήγον σήμερα, είναι πιο επίγον από το 2003. Αν ανατρέξουμε στο 2003 θα πρέπει εκεί να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους υπάρχουν τέτοιες διενέξεις στην περιοχή διότι σε τελική ανάλυση ουσιαστικά ε, αυτές είναι οι συνέπειες της εισβολής στο Ιράκ. Ε, έτσι ξεκίνησε ε, το, το όλο ζήτημα. Εμεί προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση που δημιουργήθηκε τότε στην περιοχή. Τώρα, το αποφύγουμε τον πόλεμο ε, συνεπάγεται περιορισμός, περιορισμό των στρατιωτικών δραστηριοτήτων όχι μόνο στη Συρία και στην Ιεμένη, αλλά και τον περιορισμό των πρόσφατων διανέξεων μεταξύ Ισραήλ και Ιράν στη Συριακή επικράτεια. Γι' αυτό το λόγο είναι πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση η αντιμετωπίση αυτού του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Είναι μια από τι μεγάλες απειλέ στην περιφερειακή ασφάλεια. Ο διάλογος ε, στην περιοχή είναι αυτό που θα πρέπει να επιδιώξουν οι Ευρωπαίοι, να φέρουν μαζί τις χώρες της περιοχής ε, ώστε να συζητήσουν για την ασφάλεια στην περιοχή. Το ψήφισμα του ΟΗΕ 2231 ε, που ενέκρινε τη JCTOA κάνει έκκληση για, ακριβώς γι' αυτό. Αλλά δεν μιλάμε μόνο για το Ιράν, μιλάμε και για τη Σαουδική Αραβία που εμπλέκεται στο ε, στην Ιεμένη. Να θυμίσω ότι σε παλιότερα έχει συζητήσει ε, ψηφίσματα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την απαγόρευση πώληση όπλων στη Σαουδική Αραβία. Είναι κομμάτι μια ε, συζήτηση που συνεχίζεται και σήμερα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξαρτηθεί να βρει τρόπου να φέρει του περιφερειακού παραγόντε στο ίδιο τραπέζι ώστε να περιοριστούν τέτοιε δραστηριότητε και να αποφευχθούν τέτοιε εμπόλεμε καταστάσει. Τέλο, Κάτι που ήθελα να πω ε, για τις ευρωπαϊκές δραστηριότητες. Αυτές οι δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να κατέχονται από συνοχή. Ε, γι' αυτό το λόγο συγχαίρουμε και επενούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θέλει να υπερασπιστεί την JCTOA και να διατηρήσει την εφαρμογή των διαταξιών της. Τι σημαίνει αυτό ότι ό,τι και να συμβεί στις 12 Μαΐου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ε, διέλθει από τις διατάξεις της JCTOA. Να εξετάσει οποιαδήποτε παραβίαση από οποιοδήποτε μέλος της, κοινής, ε, της Επιτροπής, ε, να αναφέρει το ζήτημα αυτό στον μηχανισμό επίλυσης περιφερειακών διαφορών, ακολουθώντας την δέουσα διαδικασία που περιγράφεται στην JCPOA όσον αφορά τέτοιου είδους παραβιάσεις. Όσον αφορά τη συνοχή και την αξιοπιστία, ε, αυτό σημαίνει συνεργασία και με το Ιράν και με τις Ηνωμένες Πολιτείες επικοδομητικά αλλά και με κριτικό τρόπο. Εγώ ανέφερα διάφορα σημεία όσον αφορά το Ιράν. Ε, συνοχή στη θεώρηση των επιθεωρήσεων της ε, ΔΟΕΑ, συνομιλίες περιφερειακές που σχετίζονται με την πυρηνική ασφάλεια, με τη μη στρατιωτική πυρηνική ενέργεια και τους πολέμους στην περιοχή φυσικά. Πολλά αναφέρθηκαν το έλλειμμα στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιράν αποτελεί ένα ζήτημα. Το Ιράν έχει την αίσθηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να εντείνει τις προσπάθειές της υπό τις παρουσίες συνθήκες και σίγουρα θα πρέπει να κάνει περισσότερα ε, εφόσον οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, ε, εγκαταλείψουν τι ε, υποχρεώσει του ε, στο πλαίσιο του JCPOA. Όσον αφορά την επικοδομητική συνεργασία με τι ΗΠΑ, παρόλα ε, στι ειδήσει που ακούμε, είναι σημαντικό οι Ευρωπαίοι να συνεργαστούν με τι Ευρωπαϊ... ΗΠΑ μέχρι τι 12 Μαΐου ώστε να βρεθεί κοινό τόπο, Οι ΗΠΑ προφανώ προφανώς δεν είναι μόνο ο προεδρό του. Θα πρέπει να γίνουν προσπάθειε λοιπόν από του ηγέτε των κρατών μελών ώστε να υπάρξουν συνομιλίε σε διάφορα επίπεδα. Αυτέ οι συνομιλίε θα είναι κάτι πολύ σημαντικό να σα ε, υπενθυμίσω ε, την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Ιράν, ε, όπου προβλέπεται μια μελλοντική στρατηγική για το Ιράν. Θυμάστε τα 4C και τα 4M. Είναι κάτι που θα πρέπει να λάβουν υπόψη η Φεντερίκα Μογκερίνη, ο Μανέλ Μακρόν, η Άγγελα Μέρκελ, ε, η Τερέζα Μέη ε, θα πρέπει να βρίσκονται, να βρεθούν στη Washington πριν από την 12η Μαΐου ώστε να συζητήσουν και να προσπαθήσουν ε, να διαβιβάσουν τις ευρωπαϊκές θέσεις. Ευρωπαϊκή θέση για μένα σημαίνει ότι θα παραμείνει αμετακίνητη στις θέσεις της όσον αφορά η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τα συμφέροντα που αναφέραμε, όχι να οδηγήσει σε κλιμάκωση, αλλά ούτε να υποχωρήσει όσον αφορά τις αρχές ε, που έχει καθιερώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το να υπάρξει μια τέτοια απόκριση αποτελεσματικά απαιτεί διερεύνηση από τα κράτη-μέλη εσωτερικά του σε ποιο βαθμό ε, σκοπεύουν να το τραβήξουν σε περίπτωση που ε, συμβεί το, αυτό, το ανεπιθύμητο στις 12 Μαΐου. Δεύτερον, τώρα τέλος, η GCPOA είναι ένα έγγραφο που έχει κυρωθεί από τον ΟΗΕ. Η Ρωσία και η Κίνα παρά τις διαφορές τους άλλα ζητήματα είναι εταίροι σε αυτής της συμφωνίας. Σε περίπτωση που το Συμβούλιο Ασφαλεία δεν καταφέρει να λάβει απόφαση σε θέματα τέτοια που αφορούν τον GCPOA, θα πρέπει να συνεργαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ω οργανισμό που μπορεί να εκπροσωπήσει την παγκόσμια κοινότητα των εθνών. Τέλος, ε, όλα όσα είπα δεν μας διασφαλίζουν την επιτυχία. Φυσικά και όχι. Αλλά ετοιμότητα, δράση, η αναγνώριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ως παράγοντα δραστήριου και ενεργού ε, θα εξαρτηθεί όχι μόνο από την επιτυχία των δρασεών της, αλλά και από την επιδίωξη μιας συνεκτικής πολιτικής με τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων, όπως θα συζητήσουμε και αργότερα και με την έβρεση ε, ε, με την αναγνώριση από όλους παράγοντες ότι έχει εργαστεί με τρόπο επικοδομητικό και συνεκτικό. Ευχαριστώ. και τώρα θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Γκέραν Μάιερ. Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ αυτούς που οργάνωσαν αυτή την ακρόση και όλους εσάς που δίδετε χρόνο για να μας ακούσετε σήμερα. Θα στοχεύσω τα σχόλιά μου για το ποια θα πρέπει να είναι η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να διατηρήσουν ε, τα κεκτημένα. Έχουμε ένα μήνα, ένα μήνα πριν ε, την απόφαση που πρόκειται να πάρει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Πρόκειται για ένα θέμα που όπως ξέρετε έχει πλήρη αρμοδιότητα και κλησική εξουσία ο Αμερικανός ε, Πρόεδρος και βεβαίως βλέπουμε ότι υπάρχουν αυτοί που τον συμβουλεύουν να παραμείνει πιστό στη συμφωνία, αλλά υπάρχουν και κάποιες αντίθετες τάσεις. Τις επόμενες εβδομάδες, όσο πλησιάζουμε δηλαδή αυτήν την ημερομηνία, πιστεύω ότι η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών θα συνεχίσει να ασκεί πίεση στους ε, τρεις, ε, τους, ε, τρεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 3 έτσι ώστε να υιοθετήσουν μια στάση που είτε θα ενισχύσει την επιβολή μονομερών κυρώσεων και θα οδηγήσει τους Ευρωπαίους να συμμορφωθούν προς αυτή τη στράση και να συνδράμουν τις Ηνωμένε Πολιτείε. Η πίεση αυτή βεβαίως, όπως ε, ξέρετε, καθορίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τους συμβούλους του Αμερικάνου Προέδρου, τα δύο νέα άτομα που τοποθετήθηκαν, οι οποίοι βεβαίως είναι σαφώς υπέρ των κυρώσεων. Θα πρέπει λοιπόν οι Ευρωπαίοι διαπραγματευτές να είναι πολύ πιο ισχυροί όσον αφορά την αντίσταση που μπορούν να προτείνουν. Όπως ξέρετε, η πιο μετριοπαθής ομάδα συμβούλων του Αμερικανού Προέδρου με τον ε, Υπουργό Εξωτερικών Τίλερσον ε, δεν είναι πια δίπλα στον Αμερικανό Πρόεδρο. Θα πρέπει λοιπόν οι Ευρωπαίοι, ο Πρόεδρος Μακρό, η Γερμανίδα Καγκελάριος και η Τερέζα Μέη, να ενισχύσουν την ε, αντίστασή τους έτσι ώστε να μετριαστεί η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών. Βεβαίως η Ευρώπη έχει λάβει αποφάσεις και σε βάση Συμβουλίου, δηλαδή 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια μπορεί να είναι λοιπόν η συλλογική αντίδραση των Ευρωπαίων. Θα πρέπει να συνεχίσει σαφώς η συζήτηση σε ανοιχτό πνεύμα με τις Ηνωμένε Πολιτείες διότι σε κάποια στιγμή θα πρέπει να συζητηθεί βεβαίως σε διάρκεια χρόνου και το θέμα της ε, λήξης της συμφωνίας. Σήμερα μιλάμε για τις ρήτρε λήξης ισχύω του ολοκληρωμένου σχεδίου, αλλά βεβαίως η συμφωνία αυτή έχει και μία ημερομηνία λήξης. Ποιες είναι οι δυνατότητες ε, αντίστασης, αν θέλετε, στο εσωτερικό αυτής της διαπραγμάτευσης και πώς μπορούμε να αξιολογήσουμε τις συνέπειες. Βλέπουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει πολύ συγκεκριμένη πολιτική και τακτική στρατηγική και σε άλλα θέματα όταν ε, συζητάμε το Κογκρέσο και διαπραγματεύεται με το Κογκρέσο και σε άλλα θέματα, μετανάστευση και άλλα και προσπαθεί να χρησιμοποιήσει πολύ συγκεκριμένη διαπραγματευτική τακτική. Το θέμα των επιπλέον μονομερών κυρώσεων που να επιβληθούν στο Ιράν καθώς και η συμφωνίες που έχουν ήδη υπογραφεί. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όσον αφορά την συγκεκριμένη συνέχεια αυτών των διαπραγματεύσεων και το τι μπορεί να συμβεί μετά τις 12 Μαΐου. Τρίτον, αυτές οι εγγύησεις από μέρους των ΗΠΑ θα πρέπει σαφώς οι Ευρωπαίοι να συνειδητοποιήσουν ότι σε κανέναν δεν θα είναι υποφελής η κατάρρευση αυτής της συμφωνίας και η κατάρρευση των σχέσεων και των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο μερών μετά την 12η Μαΐου. Θα πρέπει έτσι και αλλιώς να συνεχίσουν οι συζητήσεις και οι επαφές μεταξύ Ευρωπαίων, μέλων του Κογκρέσου και Αμερικανικής κυβέρνησης για να μετριαστούν οι αντιδράσεις και οι επιπτώσεις της κατάρρευσης αυτής της συμφωνίας. Παραδείγματος χάρη όσον αφορά την άρση και όσον αφορά τις εξαιρέξεις, τις ε, λεγόμενες ε, άλλες κατηγορίες κυρώσεων, δευτερογενείς ε, κυρώσεις, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα λαμβάνεται η απόφαση για όλα αυτά τα θέματα. Παραδείγματο χάρη η κυβέρνηση Ομπάμα, η οποία είχε μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση, πολύ πιο πολιτική της ε, όλης ε, αντιμετώπισης σε σχέση με την κυβέρνηση Τραμπ. Ένα από τα αιτήματα των Ευρωπαίων αυτή τη στιγμή είναι να μπορούν να συμμετάσχουν σε μια διαρκή βάση σε αυτή την συμφωνία. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξουν κάποιες ε, ομαδοποιήσεις διεκδικήσεων, να μπούμε δηλαδή σε περισσότερες ε, λεπτομέρειες σε κάποιες από τις ε, επιμέρους συμφωνίες. Βεβαίως υπάρχουν στρατηγικές προτεραιότητες για την Ευρώπη, όπως σας τις παρουσίασα και θα μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες και για την Ευρώπη αλλά και για το Ιράν. Ποιες είναι οι στρατηγικές προτεραιότητες. Πρώτον, για την Ευρώπη πώς μπορεί η Ευρώπη να οθήσει, να ασκήσει πίεση στο Ιράν έτσι ώστε να τηρήσει και να συμμορφωθεί με τις βασικές ε, υποχρεώσεις της σε σχέση με αυτήν την πυρηνική συμφωνία, να διατηρήσει τις δεσμεύσεις της. Δεύτερον, δεύτερη στρατηγική προτεραιότητα για τους ε, Ευρωπαίους. Εάν, εάν αποφασίσει να αποχωρήσει η Αμερικανική κυβέρνηση, θα πρέπει να μπορέσουν οι Ευρωπαίοι να υιοθετήσουν μία, αν θέλετε, συνενετική στάση, διαφορετική στάση διαφοροποίηση σε σχέση με τις Ηνωμένε Πολιτείες και όχι ε, ένα διαζύγιο με βίαιο τρόπο. Είναι πολύ σημαντικό η Ευρώπη να διατηρήσει αυτή τη στάση και είναι και πάρα πολύ δύσκολο σήμερα να μπορέσει κάποιος να προβλέψει ποια θα είναι η δράση των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι διεθνείς παρατηρητές σήμερα πιστεύουν ότι η αντίδραση του Ιράν, και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να προβλεφθεί, τους τελευταίους, ε, τις τελευταίες εβδομάδες και μέρες διαπιστώνουμε μια όξυνση, τουλάχιστον σε ρητορικό επίπεδο των, της αντίδρασης της κυβέρνησης του Ιράν. Υπάρχει απειλή ότι την επομένη της αποχώρησης των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Συμφωνία είναι σε θέση το Ιράν να εμπλουτίσει το ουράνιό του κατά 20% σε σχέση με το 5% που προβλέπεται σήμερα στη συμφωνία. Το τελευταίο χρόνο διαπιστώνουμε ότι το Ιράν παρακολουθεί πολύ στενά την ευρωπαϊκή στάση, την αντίδραση των Ευρωπαίων σε σχέση με τη δράση της Αμερικανικής κυβέρνησης και πολλές φορές έχουμε ακούσει τους Ιρανούς ηθήνοντες να επικαλούνται την εθνική ασφάλεια. Βεβαίως, σε κάθε περίπτωση το Ιράν πέρα από τη ρητορική αυτή και τις ε, καταδίκες σε λεκτικό επίπεδο πιστεύουμε ότι δεν επιθυμεί μία ραγδαία ρήξη και κατάρρευση αυτής της συμφωνίας. Αυτό θα έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις, παρόλο που υπάρχουν τα στηρίγματα από μέρους Κίνας και Ρωσίας, θα έχει πάρα πολύ σημαντικές συνέπειες για την οικονομία του Ιράν. Υπάρχουν λοιπόν αρκετά κίνητρα για την κυβέρνηση του Ιράν, έτσι ώστε να παραμείνει εν μέρη τουλάχιστον ε, δεσμευμένη σε σχέση με τη συμφωνία αυτή βλέπουμε ότι είναι πλέον ε, σαφές για τους Ιρανούς, για τους Ιρανούς πολίτες, για την ε, κοινή γνώμη στο Ιράν, ότι αυτή η συμφωνία έχει ε, ωφέλη και θετικές επιπτώσεις και οικονομικές, αλλά και για την ασφάλεια του Ιράν. Πιστεύουμε λοιπόν ότι σε κάποια μορφή θα συνεχίσουν οι δεσμεύσεις του Ιράν, οι διαπραγματεύσεις και θα πρέπει να αναρωτηθούμε αν οι Ευρωπαίοι θα είναι σε θέση να προτείνουν ένα μηχανισμό, μια διαδικασία έτσι ώστε να αντισταθούν στις επιπτώσεις ε, σε περίπτωση που η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών αποφασίσει για την ε, πάυση της άρσης των κυρώσεων όσον αφορά βεβαίως συγκεκριμένα τις επιπτώσεις αυτές επί των ε, ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Αν αποχωρήσει η Αμερική, θα πρέπει καταρχήν η ε3 να δημιουργήσουν μια μεγαλύτερη συμμαχία έτσι ώστε να υπάρξει πιο αποτελεσματική αντίδραση στην απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αυτό βεβαίως εισπυρώνοντας τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενσωματώνοντάς τους στις συζητήσεις, στις διαπραγματεύσεις, αλλά και κάτι παραπάνω. Βεβαίως ε, και η Ρωσία, η Ινδία η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία, όλη η Ασία η οποία πλήττεται από την κατάρρευση μιας τέτοιας συμφωνίας. Οι επιπτώσεις για τη Μέση Ανατολή είναι γνωστές, ανησυχούν όλοι και για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, ιδιαίτερα αν συνεχίσουν να επιβάλλονται αμερικανικές κυρώσεις μονομερός. Και βεβαίως και για το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και για τις ε, πολύ σημαντικές ε, ευρωπαϊκές οικονομίες οι επιπτώσεις θα είναι άμεσες. Θα πρέπει λοιπόν να παρακολουθήσουν οι ευρωπαϊκές χώρες, οι ευρωπαϊκές οικονομίες, ποιες θα είναι ακριβώς οι αποφάσεις που θα λάβει η Αμερικανική κυβέρνηση, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις επί ε, ευρωπαϊκής οικονομίας, των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Σίγουρα οι επιπτώσεις και τα συμφέροντα των Ευρωπαίων θα πληγούν και αυτό θα πρέπει να παρακολουθεί πολύ στενά. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αλλά και ο ιδιωτικός τομέας θα πρέπει να εξετάσει όλες τις περιπτώσεις εξαιρέσεων για ευρωπαϊκές εταιρείες ή για ευρωπαϊκούς τομείς και θα πρέπει να εξουδετερωθούν στο ελάχιστο οι επιπτώσεις αυτές. Παραδείγματο χάρη, οι τομεί, όπως ο, τραπεζο, ο τραπεζικός χρηματοπιστωτικός, οι αεροπορικές μεταφορές, η ενέργεια θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξαιρεθούν, να διαπραγματευτούν δηλαδή με το Κογκρέσο οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις συγκεκριμένες εξαιρέσεις για κάποιους τομείς ιδιαίτερα σημαντικούς για την ευρωπαϊκή οικονομία. Ξέρω ότι αυτό που σας λέω δεν είναι κάτι που εύκολα θα συμφωνήσουν οι Βρυξέλλες, αλλά υπάρχουν και οι λεγόμενες ε, ρήτρες και κανόνες παρεμπόδισης της Ευρώπης η αναζωγόνηση αυτών των κανόνων παρεμπόδισης από μέρους της Ευρώπης, blocking regulation, είναι επίσης κάτι που θα πρέπει σοβαρά να μας απασχολήσει. Και ξέρω ότι αυτοί οι κανόνες παρεμπόδισης από μέρους της Ευρώπης είναι κάτι που δεν είναι εύκολο να ενεργοποιηθεί, αλλά έχω μιλήσει με πολλούς εκπροσώπους πολυεθνικών ε, επιχειρήσεων και ομίλων και ξέρω ότι σίγουρα αυτοί οι κανόνες παρεμπόδισης της Ευρώπης μπορεί να έχουν κάποια αποτελέσματα και σε πολιτικό επίπεδο. Αλλά αυτό σε συνδυασμό με μια πολύ συγκεκριμένη διαπραγμάτευση κάποιων εξαιρέσεων για τομείς ε, συγκεκριμένους που είναι ε, ουσιαστικοί για την ευρωπαϊκή οικονομία. Ξέρω ότι η ευρωπαϊκή κυβέρνηση επεξεργάζεται ήδη το θέμα του τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού τομέα. Σαφώς η συμφωνία αυτή θα έχει επιπτώσεις στον τομέα αυτό και υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο παράρτημα της συμφωνίας που αναφέρεται στον τραπεζικό τομέα καθώς και τις επιπτώσεις και για το Ιράν αλλά και για τις ευρωπαϊκές ε, οικονομίες. Προβλέπει η συμφωνία σημαντικές μεταρρυθμίσεις και δεσμεύσεις από μέρος του Ιράν για αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο τραπεζικό του σύστημα. Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στον τομέα αυτό από μέρος του Ιράν δεν είναι εντυπωσιακή. Οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στο Ιράν τις τελευταίες δεκαετίες βεβαίως παρόλο που η άρση τους έλαβε χώρα το 2016, έχουν οδηγήσει τον τραπεζικό τομέα του Ιράν σε ένα τέλμα. Ε, ένα άλλο σημείο είναι ότι θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή η δυνατότητα διαπραγμάτευσης με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Η... Τα εμπλεκόμενα μέρη σίγουρα μπορεί και εκεί να προχωρήσουν τις συζητήσεις που έχουν ήδη ξεκινήσει σύσταση που θα ήθελα να σας υποβάλω προς είναι ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε και άλλους εταίρους σε αυτή την υπόθεση όπως η Σαουδική Αραβία, το Ισραήλ. Δεν πρέπει οι Ηνωμένε Πολιτείε να ξεχνούν ότι πρόκειται για ένα θέμα εθνικής ασφάλειας, πρόκειται για θέμα πυρηνικής ασφάλειας σε μια περιοχή στην Μέση Ανατολή, πολύ κοντά στην Ευρώπη και σίγουρα οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να παίξουν ένα καθοριστικό ρόλο γιατί είναι οι πρώτοι που θα πληγούν εάν υπάρξει κλιμάκωση. Ευχαριστώ πολύ. Θα γίνει συζήτηση. Θα πρέπει να δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Λίτς που θα μιλήσει εξ ονόματος του κυρίου Φλέκενστάιν που είναι ο αρμόδιος ε, ε, από την Επιτροπή μας για τις σχέσεις με το Ιράν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, επίσης ευχαριστώ πολύ για αυτές τις δύο ε, βαθιές ε, περιγραφές που μας δώσετε. Μιλώ εξ ονόματος του Κουρτ Φλέκενστάιν που κολλείται και απουσιάζει σήμερα, αλλά σας στέλνει χαιρετισμού. Και υποστηρίζω και εγώ αυτά που λέει. Ως ε, εισηγητής για το Ιράν, λέει ο κύριος Φλέκενστάιν, θέλω να τονίσω τη σημασία της σημερινής δημόσιας ακρόασης για την εγώμενη ε, συμφωνία με το Iran GCPOA και είναι πάρα πολύ σημαντικό να συζητήσουμε τις ε, δυνατότητες επιλογής και πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση της αποχώρησης των Πολιτειών. Η συμφωνία του Ιράν ε, είναι θέμα ασφαλείας για τη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη και τον κόσμο ολόκληρο. Η καταστροφή αυτής της συμφωνίας θα υπονομεύσει τους μετριοπαθείς στο Ιράν που υποστηρίζουν τη συμφωνία. Αν ε, κρατήσουν οι σκληροπυρηνικοί θα επανέλθει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν αλλά και η συγκρουσιακή του στάση στην περιοχή όπως και οι δύο είπατε. Γι' αυτό συμφωνώ απολύτως με την είπατε εκπρόσωπο όταν τόνισε τη στρατηγική σημασία ε, που έχει η πλήρης ε, υλοποίηση της συμφωνίας από όλα τα μέρη στην Υπουργική Συνάντηση την περασμένη εβδομάδα. Μέχρι τώρα οι διεθνείς... Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας επανειλημμένα έχει τονίσει και έχει επαληθεύσει ε, ότι ε, ε, τα τηρεί όλα αυτά το Ιράν. Μετά τους νέους διορισμούς του Μάικ Πομπέα και άλλων στις Ηνωμένε Πολιτείε αυξάνεται ο κίνδυνος να ανατραπεί η συμφωνία το Μάιο η ε, κυβέρνηση Τραμπ ε, δείχνει πιο σκληρή στάση για την πυρηνική αυτή συμφωνία. Γι' αυτό θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι έχουμε και στρατηγικές προτεραιότητες και προθεσμίες και παραμένουμε προσιλωμένοι στην τήρηση της συμφωνίας. Βεβαίως, χρειάζεται κοινή προσπάθεια από τις διάφορες πλευρές συμφωνίας έτσι ώστε να τηρείται η πλήρης εφαρμογή. Αλλά βασικό μας συμφέρον είναι να παραμείνει το Ιράν ε, στην πλήρη συμμόρφωση με τη συμφωνία αυτή, αλλά και οι Ηνωμένε Πολιτείε να παραμείνουν προσιλωμένε στην επιτυχία αυτή τη συμφωνία. Στην Ευρώπη χρειάζεται δράση, ενότητα και κοινή στόχη. Χρειάζεται να διατρανώσουμε περισσότερο τη θέση μα στι επόμενε συνομιλίε προ τι Ηνωμένε Πολιτείε, για να μην γίνουμε συνένοχοι στην υπονόμευση της πυρηνικής συμφωνίας. Είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε ότι θέλουμε να ε, δούμε εναλλακτικού τρόπους διαφύλαξης αυτής της συμφωνία σε περίπτωση που υποχρεωθούμε να το κάνουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι και θα συνεργαστούμε με ε, ομονοούντες συμμάχους για να ε, παρακάψουμε την αποχώρηση ε, των ΗΠΑ. Αλλιώς θα αυξηθεί ο κίνδυνος σύγκρουσης και περισσότερων σειράξεων στην περιοχή και το κόστος βασικά θα το πληρώσει μάλλον η Ευρώπη. Θα πρέπει να εξακολουθήσουμε να δείχνουμε ότι η Ευρώπη είναι αξιόπιστος εταίρος και θέλει να τηρείται το διεθνές δίκαιο σε δύσκολους καιρού. Βεβαίω είμαστε πάντα πρόθυμοι να συζητήσουμε και άλλα θέματα με το Ιράν, εκτός της πυρηνική συμφωνίας και του πεδίου εφαρμογή δύο διαφορές που έχουμε για το βαλιστικό πρόγραμμα ε, και τις εντάσεις στην περιοχή η Συρία και η Εμένη. Όλα αυτά είναι βεβαίως παρόντα θέματα, αλλά είναι ξεχωριστά και θα πρέπει να ειδωθούν εκτό τη συμφωνία. Και τέλο, χωρί αυτό είναι το λιγότερο σημαντικό, θα πρέπει να προετοιμαστούμε για το χειρότερο σενάριο ε, τη αποχώρηση των ΗΠΑ και επιβολή κυρώσεων από πλευρά του στο Μάιο. Θα πρέπει να δώσουμε πολιτικά και οικονομικά κίνητρα στο Ιράν για να μπορεί να συνεχίσει να εφαρμόζει τη συμφωνία. Συζητούμε ποιες είναι αυτές οι δράσεις ε, με πολιτικά και τεχνικά μέσα για να προστατεύσουμε και τις ευρωπαϊκές εταιρείες από δευτερογενείς κυρώσεις. Ανταλλαγές απόψεων σε ακροάσεις όπως αυτή θα βοηθήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να περιορίσει τις ζημίες. Και θα ήθελα εδώ να προσθέσω και κάτι ακόμα, πέρα από το όσα είπε ο κύριος Φλέκενστάιν, ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε και άλλα στρατηγικά ζητήματα στην περιοχή. Υπάρχει κάποιο ευρωπαϊκό κράτος που εκτρέπεται. Και τι θα μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με αυτό. Μιλήσατε για περιφερειακές συνομιλίες. Θα πρέπει να δούμε και τα πυρηνικά γενικότερα στο Περσικό κόλπο. Γίνονται συνομιλίες. Εσείς αναφερθήκατε στη Σαουδική Αραβία. Αυτά λαμβάνονται ήδη υπόψη. Παράλληλα δηλαδή ένας άλλος δρόμος πέρα από το πρόγραμμα και τη συμφωνία η κατάσταση είναι πάρα πολύ τεταμένη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Τάνοκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα πρέπει να φύγω γρήγορα, παρακαλώ, αν μου απαντήσετε πρώτον. Συμφωνώ φυσικά με τις ανησυχίες για τις πρόσφατες ε, ε, εξελίξεις και το διορισμό του Συμβούλου αυτού που είναι διαβόητος ε, αντίπαλος του Ιράν. Εδώ έχει προτείνει στρατιωτική προληπτική δράση. Και πραγματικά υπάρχει κίνδυνο οι Ηνωμένε Πολιτείε να αποσυρθούν από τη συμφωνία με το Ιράν. Δύο γρήγορε ερωτήσει. Κάποιο από του ομιλητέ είπε ε, ότι το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας είχε προσυπογράψει ε, τη συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών. Δεν το ήξερα. Ισχύει κάτι τέτοιο. Πραγματικά σωστά σας κατάλαβα. Έχουν προσχωρήσει στη συνθήκη μη διάδοσης και πώς θα κάνουν πυρηνικά με ή χωρίς συμφωνία ε, πυρηνικών για το Ιράν, χωρίς ε, να ε, υποστούν κυρώσει από το ΝΟΙΕ. Γιατί αν είσαι μέρο της συμφωνίας μη διάδοση δεν μπορείς να αναπτύσσει πυρηνικά. Ε, δεύτερον, η ίδια μου η χώρα σε ένα χρόνο θα φύγει. Είναι μέλο του Συμβουλίου Ασφαλείας βεβαίως και μέρος των κρατών που διαπραγματεύονται Τρει. Το Ηνωμένο Βασίλειο πραγματικά αγωνιά να ε, έχει μια εμπορική συμφωνία με τις Ηνωμένε Πολιτείε ε, για το 20 μήνο μετά το Brexit, τη μεταβατική αυτή περίοδο. Και μάλλον οι ε, Ηνωμένε Πολιτείε το βλέπουν με κάποιο καχύποπτο πνεύμα λόγω προστατευτισμού. Αλλά υπάρχει αυτό το αγγλοσαξονικό μέτωπο ε, και εμπορικά είμαστε πιο πολύ συνδεδεμένοι και στραμμένοι με τις Ηνωμένε Πολιτείε μετά το Brexit. Πώς μπορεί λοιπόν το Ηνωμένο Βασίλειο πλέον εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρόλο που λέει ότι θέλει να υποστηρίξει το σχέδιο δράσης ε, GCPOA ως τρίτη χώρα, Πώ θα τετραγωνίσει τον κύκλο το Ηνωμένο Βασίλειο ε, σε ό,τι αφορά τι δευτερογενεί κυρώσει. Αυτό είναι πραγματικό δίλημα για το Λονδίνο ουσιαστικά. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μούντι. Thank Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις και όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε. Συμφωνώ πρώτα απ' όλα με τα σχόλια που ακούσαμε όσον αφορά το JCPOA και το πού βρισκόμαστε και την υποστήριξη της συνέχισης αυτής ε, της διαδικασίας και το πόσο σημαντικό είναι να διατηρηθεί το δίκαιο ε, στο πλαίσιο των διεθνών μας ε, συμφωνιών. Πρέπει να τηρήσουμε τις συμφωνίες αυτές και τις ευθύνες μας. Είναι πολύ σημαντικό. Ένα από τα πράγματα που αναφέρατε και θα ήθελα να το αναλύσετε λίγο παραπάνω είναι το σημείο που αφορά τις δράσεις κατά του Ιράν εκτός του JCPOA διότι αναμφίβολα εκφράζονται αμφιβολίες ε, για το Ιράν και για τα όσα συμβαίνουν εκεί όσον αφορά το λαό του Ιράν αλλά και τους λίπους λαούς ε, ε, αλλά και ανθρώπους που έχουν φυλακιστεί είναι, δεν είναι παρά ένα παράδειγμα των όσων συμβαίνουν εκεί και επίσης και γίνονται και κάποιες συζητήσεις σε σχέση επιπλέον ε, κυρώσεις ε, πέραν του JCPOA. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, σε, έχουμε και τη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών ε, σε σχέση με την JCPOA και δράσεις που είναι πιθανώς να εφαρμοστούν σε σχέση με τα όσα γίνονται εντός του Ιράν και που σχετίζονται ή δεν σχετίζονται με την πυρηνική συμφωνία. Δεύτερον, όπως έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη. Διάφοροι ε, κατεξουσιοδότηση πόλεμοι που συμβαίνουν ε, στην περιοχή. Και το ερώτημα είναι, ε, έχουν ξεκινήσει ήδη περιφερειακές συνομιλίες σε σχέση με όλα αυτά. Από τα όσα είπατε δεν κατάλαβα πολύ καλά. Επιστέτε μια νέα JCPOA που να αφορά την κατάσταση της Σαουδική Αραβία. Τι ακριβώς θέλετε σε σχέση με αυτή την εξέλιξη. Θα παραμείνω σε αυτές τις δύο ερωτήσεις. Είναι πολύ ευαίσθητη η κατάσταση Ε, τα πράγματα είναι πολύ πιο επικίνδυνα σε σχέση, από, σε με την εποχή που ξεκινήσαμε τις συζητήσεις για την JCPOA. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στους χειρισμούς μας στο άμεσο μέλλον. Ευχαριστώ. Ο Τάκης παρακαλώ. Σας ευχαριστώ και εγώ για τις εξαιρετικές σας παρουσιάσεις. Δύο ερωτήσεις έχω. Μία για τον κύριο Κονέλιος Άντεμπα. Είπατε ότι μέχρι τα τέλη της συμφωνίας το Ιράν θα έχει μεταμορφωθεί, θα είναι μια διαφορετική χώρα. Δεν ξέρω αν το κατάλαβα απολύτω και θα ήθελα παρακαλώ να το αναλύσετε περισσότερο. Και για την κυρία Γκέραν Μαγέ. Είπατε ότι η οικονομία σε κάποιες χώρες θα επηρεαστεί αρνητικά ε, λόγω της συμφωνίας και εννοείται την Ινδία, την Νότια Κορέα κλπ. Αυτό δεν το κατάλαβα πάρα πολύ καλά. Και στη συνέχεια αναφερθήκατε στην τακτική που χρησιμοποίησε ο κύριος Τραμπ όταν διαπραγματευόταν με το Κογκρέσο. Και είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να τα, λάβει όλα αυτά ή να τα λάβει υπόψη της. Τι ακριβώς εννοείται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής. Θα ήθελα κι εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ ε, για την καλή παρουσίαση, λέει ο κύριος Βούχνερ. Έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση, η οποία επιμένει ε, σε ένα θέμα που αναφέρθηκε επανειλημμένα. Πώς θα αντιδράσει η Ευρώπη εάν έρθει το χειρότερο σενάριο και αποσυρθούν οι Ηνωμένε Πολιτείε από τη συμφωνία και επιβάλλουν ε, δευτερογενείς κυρώσεις για τις ευρωπαϊκές εταιρείες. Θεωρώ ότι δεν θα υπάρχει δυνατότητα παράκαμψη ή αποτροπή των δευτερογενών κυρώσεων, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο μέρο του. Το χρηματοπιστωτικό τομέα το βλέπουμε ήδη από τώρα. Επηρεάζονται ε, οι εταιρείε μα. Ερώτηση. Πιστεύετε πραγματικά ότι η Ευρώπη είναι αρκετά ισχυρή έτσι ώστε να αντισταθεί και να επιβληθεί κατά των δευτερογερών ακυρώσεων τον είπα. Ερώτηση δεύτερη. Πώς εκτιμάτε την κατάσταση ιδιαίτερα σε σχέση με τη Βόρεια Κορέα. Εδώ και καιρό υπάρχει καλή συνεργασία μεταξύ Ιράν και Βόρειας Κορέας, τουλάχιστον σε τούτο εδώ το κομμάτι. Αν εμείς τώρα εδώ ε, απαιτήσουμε διάφορα πράγματα από τη συμφωνία και επιβάλλει και την άποψή του ο Τραμπ για το βαλιστικό, το πυραυλικό ε, πρόγραμμα του Ιράν, αν μειωθεί, βοηθάει πραγματικά αυτό. Γιατί το Ιράν πατάει και ένα πόδι στη Βόρεια Κορέα και μπορεί να πάρει από εκεί διάφορα υλικά που χρειάζεται ή που θέλει. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φρόιντς. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρετε, όταν είναι κανεί τελευταίο στη σειρά των ομιλητών, τότε οι περισσότερε ερωτήσει έχουν ήδη γίνει. Άκουσα τον κύριο Μπούχνερ μόλι τώρα, ο οποίο έκανε αυτό το ερώτημα για τη Βόρεια Κορέα. Και χαίρομαι. Χαιρόμουν εγώ που είχα αυτή την ερώτηση στα χέρια μου που κανεί δεν είχε κάνει πριν, αλλά έμεινε και κάτι και για μένα από το ερώτημα της ε, Βόρειας Κορέα που έθεσε ο κύριος ε, Μπουχνέρ. Κάτι που ξέχασε. Ε, λίγο διαφορετικό από αυτό που έθεσε ο κύριος Μπουχνέρ. Κατά την άποψή σας, σε περίπτωση που υπάρξουν διαπραγματεύσεις μεταξύ του κυρίου Τραμπ ε, και του Κιμ Ιωμούν, πώς θεωρείτε ότι τέτοιες διαπραγματεύσεις θα επηρεαστούν από οτιδήποτε κάνει ο Τραμπ, γιατί δεν ξέρουμε τι θα κάνει στις 12 Μαΐου. Σε περίπτωση όμως που ε, αποσυρθεί από την JCPOA, τι θα σημάνει αυτό, τι μήνυμα θα είναι αυτό προς τη Βόρεια Κορέα σε περίπτωση διαπραγμάτευσης παρόμοια συμφωνίας από τον Τραμπ. Διότι παρόμοια θα πρέπει να είναι η συμφωνία διότι είναι σχετικά τα ζητήματα αυτά μεταξύ του. Σε περίπτωση λοιπόν που θέλει να διαπραγματευτεί κάτι τέτοιο Τραμπ με τη Βόρεια Κορέα, Πώ θα επηρεαστεί αυτή η διαπραγμάτευση. Να δω αν έχω κάτι άλλο να ρωτήσω. Όχι, νομίζω όλα ρωτήθηκαν. Ακόμη και το ερώτημα που έθεσε ο κ. Χατζηγεωργίου, το διαφορετική χώρα, τι εννοείται, πώ εννοείται ότι θα είναι διαφορετικό το Ιράν στο τέλο τη συμφωνία από αυτό που ξεκίνησε τη διαπραγμάτευση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, απάντηση με τη σειρά που θέλετε. Όποιος από τους δύο. Thank you. Uh, thank you. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ και τα μέλη ε, που επιμένουν ε, στις ερωτήσεις για να δούμε τα θέματα σε μεγαλύτερο βάθος. Θα απαντήσω στις ερωτήσεις που κάνατε σε μένα ή σε κάποιες γενικές και μετά θα απαντήσει συνάδελφος σε υπολοιπα Το πρώτο, αυτό που ρώτησε ο Άρνε ε, για τα αποκλεινόμενα συμφέροντα των κρατών μελών. Εσείς θα γνωρίζετε αυτά καλύτερα από μένα. τα αποκλίνοντα μάλλον, και τι ε, πολιτική έχει ο καθένας απέναντι στο Ιράν. Δημοσιεύματα φέρουν τους τρεις Ευρωπαίους, ε, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Γερμανία, να πήγαινε προς την ίδια κατεύθυνση αλλά ε, ε, και κάποιες διαφωνίες μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών. Ε, αυτό δεν είναι τίποτα το καινούριο, γιατί ε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο ε, τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 12 χρόνια μέχρι το 2015 και τη συμφωνία να συμφωνήσουν μεταξύ τους οι ευρωπαϊκές χώρες ακριβώς γιατί υπάρχει διαφορετικότητα και ποικιλία στην ευρωπαϊκή προσέγγιση. Ε, Παρ' όλα αυτά χρόνο δεν έχουμε μέχρι το Μάιο ε, για να αναλωνόμαστε σε συζητήσεις για αυτά τα θέματα και τα ε, αποκλείοντα συμφέροντα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει θέση. Μπορεί να είναι η θέση των τριών αυτών κρατών, αλλά χρειάζεται κάποια κοινή θέση. Ε, οι περιφερειακές συνομιλίες δεν έχουν αρχίσει ακόμα. Αναφέρθηκαν, έγινε μια πρόταση, όπως σας είπα προηγουμένως, από το ίδιο το Ιράν, που είναι πρόθυμο να ε, μπει σε περιφερειακές συνομιλίες. Η Σαουδική Αραβία ε, είναι διστακτική και επιφυλακτική να μπει σε συνομιλίες για την περιφερειακή ασφάλεια. Το θέμα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση τι θα κάνει και τα μεμονωμένα κράτη-μέλη της. Μπορούν να αναγκάσουν το ΡΙΑΤ να μπει σε τέτοιες συνομιλίες. Πάντως το πνεύμα της συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ακριβώς η αναζήτηση πολυμερών λύσεων σε τέτοιου είδους συγκρούσεις. Και κατά τα άλλα, καλό θα ήταν να δεχτούμε τουλάχιστον την προσφορά των Ιρανών και να αρχίσουν περιφερειακές συνομιλίες. Με ρωτήσατε σε ποιο βαθμό το Ιράν θα είναι διαφορετική χώρα μέχρι το 2031. Γιατί για τέτοιο ορίζοντα μιλούμε 15 ετίας μετά τη συμφωνία. Ο καθένα μπορεί να τρέφει διάφορες ελπίδες για το πώς θα είναι τότε το Ιράν, αλλά εγώ δεν ήρθα εδώ για να καλλιεργήσω ελπίδες. Αυτό που εννοώ είναι ότι και μόνο η τεχνική και η νομική κατάσταση, το πλαίσιο θα είναι διαφορετικό εάν εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία όπως είχε σχεδιαστεί. Μετά από μία οκταετία ε, ζήτησε το Ιράν να επικυρώσει το συμπληρωματικό πρωτόκολλο. Μέχρι τώρα είναι εθελοντική εφαρμογή του. Η επικύρωση του συμπληρωματικού πρωτοκόλλου συνδέεται προφανώς με ε, την έναρξη ε, νομικής διαδικασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες για να αρθούν οι κυρώσεις, πράγμα πίθανο αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά η συμφωνία έχει την εξή κεντρική ιδέα, ότι ε, το Ιράν δεν θα είναι στο status quo ante σε αυτό που επικρατούσε πριν τη συμφωνία, όταν λήξει η συμφωνία αυτή. Αυτό εννοούσα. τώρα, μια άλλη ερώτηση. Α, ζητώ συγγνώμη. Κύριε Τάνοκ, έφυγε ο κύριο Τάνοκ, αλλά η Σαουδική Αραβία βεβαίω έχει υπογράψει τη συνθήκη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων. Και βεβαίω δεν επιτρέπεται να αναπτύξει πυρηνικά όπλα, αλλά ε, έχει δηλώσει και έχει απειλήσει δημόσια ότι θα το κάνει εάν ε, το κάνει το Ιράν. είναι πολύ λίγα τα μέλη της Συμφωνίας Μη Διάδοσης των Πυρηνικών που συζητούν τέτοια δυνατότητα να αναπτύξουν πυρηνικά. Η Σαουδική Αραβία θα πρέπει να αποσυρθεί από τη συμφωνία αυτή, όπως έκανε και η Βόρεια Κορέα. Και γενικά θα υποστεί τις ίδιες κυρώσεις με τη Βόρεια Κορέα και με το Ιράν, όταν υπήρξε υποψία ότι αναπτύσσει πυρηνικά όπλα. Αυτό δεν θα πρέπει να το ε, κοιτάζουμε επιπόλαια για ψήφιση, αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μηχανισμός να, ε, να φτιάξει πυρηνικά η Σαουδική Αραβία, όντας μέλος της συνθήκης μη διάδοσης. Έγινε μια ερώτηση για το πώς θα αντιδράσει η Ευρώπη ενδεχομένω. και πώς θα αντιταχθεί στις δευτερογενείς κυρώσεις των ΗΠΑ. Εδώ εμεί δεν οικοτολογούμε για το τι είναι πρόθυμη ή τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε, να δώσουμε δωσουμε καποιε συμβουλέ για το πώ θα διαμορφωθεί η Ευρωπαϊκή θέση. Έκανε κάποια σχόλια η Έλλη. Ε, τι θα μπορούσε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση αν είχε κοινή θέση για να αντιμετωπίσει τι δευτερογενείς κυρώσει. Αλλά και πάλι το ερώτημα εν μέρη μόνο έχει να κάνει με το αν θα είναι αποτελεσματικές αυτές οι ασφαλιστικές δικλείδες. Το θέμα είναι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την προθυμία να, να πάει προς μια κατεύθυνση ενόψει της 12ης Μαΐου. Αυτή τη στιγμή ε, την η Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάποιες δηλώσεις, σε κάποιες ε, ε, επιθέσεις ε, στις ε, απόψεις κάποιων άλλων, αλλά δεν υπάρχει η ίδια η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τι προτίθεται να κάνει στη χειρότερη περίπτωση. Και δεν είναι μόνο χειρότερη περίπτωση, αλλά είναι για να έχει θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα γενικότερα ζητήματα και πώς ε, αντιμετωπίζει τα γενικότερα περιφερειακά ζητήματα, ζητήματα ασφαλείας και άλλα. θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρουσιάσει μια συνολική πρόταση, ένα πακέτο ας πούμε για την περιοχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ε, κυρία Κεράν μαγιά. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω και εγώ να απαντήσω τα σημεία στα οποία δεν απάντησε ο συνάδελφος. Όσον αφορά την ευρωπαϊκή σχέση, καθώς ε, και τις δραστηριότητες ε, οι οποίες δεν άπτονται του πυρηνικού τομέα και τη στάση του Τραμπ. Καταρχήν, οι νέες κυρώσεις που μπορεί να επιβληθούν εκ νέου στο Ιράν θα έχουν σίγουρα επιπτώσεις και βεβαίως εδώ θα συμπεριλάβω και το θέμα των βαλιστικών πυράβλων, εκτός των πυρηνικών. Υπάρχουν πολλά επίμαχα, αν θέλετε, σημεία μεταξύ Ιράν και των άλλων μέρων της συμφωνίας και σαφώς δεν είναι οι κυρώσεις ε, αποκλειστικά και μόνο το μόνο όπλο που μπορεί να έχουμε. Το θέμα τώρα των ε, πυραυλικών προγραμμάτων του Ιράν και των προτεραιοτήτων, των στρατηγικών προτεραιοτήτων το πώς κάποιος μπορεί να ταξινομήσει, αν θέλετε, τα διάφορα προβλήματα, τα διάφορα επίμαχα σημεία που μπορεί να έχουμε στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και πώς μπορεί να αντιμετωπίσει τους ε, επιμέρους αυτούς τομείς. Είδαμε ότι σαφώς οι κυρώσεις δεν είχαν πάντα τις ε, συνέπειες και τις επιπτώσεις που περιμέναμε. Σαφώς λοιπόν σε κάποιους τομείς οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν είχαν αποτελέσματα, σε κάποιους όχι. Το θέμα είναι και ο χρόνος, αλλά και το πόσο αυτές οι κυρώσεις πραγματικά έπληξαν τομείς. Γι' αυτό και σήμερα κοιτάμε πώς μπορεί η δράση να κατανεμηθεί διαφορετικά έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί το αποτέλεσμά τους. Και νομίζω ότι η κυβέρνηση Τραμπ το έχει αντιμετωπίσει αυτό. Οι αντίπαλοι της συμφωνίας στο εσωτερικό της κυβέρνησης Τραμπ αλλά και οι σύμβουλοι Τραμπ οι οποίοι είναι κατά της συμφωνίας αντιμετωπίζουν και αυτές τις συνέπειες και την αποτελεσματικότητά τους θέλουν κατά κάποιο τρόπο η συμφωνία να παραμείνει και να οδηγήσουν και τους Ευρωπαίους αλλά και την Αμερικανική κυβέρνηση σε μία όξυνση της τάσης τους έτσι ώστε να μην μπορέσει πλέον το Ιράν να δεσμεύεται στην αρχική συμφωνία, να τους αναγκάσουν δηλαδή να βγουν από τη συμφωνία. Αν λοιπόν εμείς αποφασίσουμε να πάρουμε κάποια απόφαση. Αν δηλαδή οι Ευρωπαίοι αποφασίσουν πραγματικά να ακολουθήσουν τις ΗΠΑ και να βγουν εκτός συμφωνίας, θα πρέπει σίγουρα να δείξουμε στους ε, Ιρανούς ότι θέλουμε να παραμείνει η συμφωνία ζωντανή. Δεσμευόμαστε για τη συμφωνία, αλλά την ίδια ώρα θέλουμε να σας δείξουμε ότι και το Ιράν πρέπει να δεσμεύεται και το Ιράν πρέπει να παραμείνει πιστό. Υπάρχει ένας τεράστιος βαθμός απροβλεψιμότητας, αν θέλετε, όσον αφορά την αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών. Βλέπουμε ότι και από ρητορική απόψεως, αλλά και από απόψεως στρατηγικής, οι Ηνωμένε Πολιτείε σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολο να προβλέψουμε την μελλοντική του στάση και δράση. Μου κάνατε και μία ερώτηση για τις επιπτώσεις στην οικονομία, την Ασιατική, Ινδία, Ιαπωνία. Υπάρχουν διαπραγματεύσεις για μεγάλες συμφωνίες με το Ιράν. Σαφώς και έχουν κάθε συμφέρον όλες αυτές οι χώρες στην Ασία να υπάρξει αποκλιμάκωση να μειωθεί η ένταση στην περιοχή και σίγουρα θα χαιρετήσουν με πολύ θετικό τρόπο ένα συντονισμό με την ευρωπαϊκή στάση. Και σίγουρα το μήνυμα της αποχώρησης των Ηνωμένων Πολιτειών από τη συμφωνία, η κατάρρευση της συμφωνίας σίγουρα θα είναι ένα πάρα πολύ αρνητικό μήνυμα για την Ασία. Βεβαίως και η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει την θέση της, τη φωνή της. Βεβαίως και το Ηνωμένο Βασίλειο, βεβαίως και οι μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες ε, είναι ένας καθοριστικός παράγοντας για το Ηνωμένο Βασίλειο στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα σίγουρα ο τομέας αυτός είναι πάρα πολύ σημαντικός και πιστεύω ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να παραμείνει κοντά στην Ευρώπη, κοντά στους ευρωπαϊκούς ε, εταίρους. Όσον αφορά βεβαίως το τεχνικό κομμάτι αυτής της συμφωνίας, θα πρέπει να παραμείνουμε δεσμευμένοι και κοντά στις ευρωπαϊκές θέσεις. Πιστεύω, αναφερθήκατε στη Σαουδική Αραβία, Βεβαίως και υπάρχουν σε περιφερειακό επίπεδο διαπραγματεύσεις, συζητήσεις με το Ιράν. Ο τελευταίος γύρος διαπραγματεύσεων που έλαβε χώρα πολύ πρόσφατα τον Ιανουάριο στην συνάντηση υψηλού επίπεδου στο Μόναχο για θέματα εθνικής ασφάλειας. Εκεί συζητήθηκε σοβαρά και ο ρόλος της Σαουδικής Αραβίας, η εμπλοκή τους ε, στην Ιεμένη η όπλων από μέρους των ευρωπαϊκών χωρών και βεβαίως όλη η προσπάθεια να εξουδετερωθεί, να μετριαστεί η ένταση, η κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή θα πρέπει να συνεχιστούν. Μία τέτοια, αν θέλετε, αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών και κατάρρευση συμφωνία σίγουρα θα εντείνει την κατάσταση. Και η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη, το Ισραήλ το ΡΙΑΝΤ σίγουρα μπορεί να παίξουν ένα καθοριστικό ρόλο σε αυτήν την προσπάθεια δημιουργίας ενός μηχανισμού αποκλιμάκωσης της έντας στην περιοχή. Ε, θα απαντήσω και στην ερώτηση για τη Βόρεια Κορέα. Εδώ υπάρχουν διστάμενες απόψεις μεταξύ μας. Αλλά εγώ πιστεύω ότι η πυρηνική ασφάλεια και όσοι ασχολούνται με αυτήν σίγουρα θεωρούν ότι μία κατάρρευση αυτής της συμφωνίας με το Ιράν σίγουρα θα υπονομεύσει την αξιοπιστία μιας μελλοντικής πιθανής συμφωνίας με τη Βόρεια Κορέα για παρόμοια θέματα. Πώς μπορεί η Αμερικανική κυβέρνηση με αξιοπιστία να ισχυρίζεται ότι θέλει να συνάψει συμφωνία και να προχωρήσει σε σοβαρές διαπραγματεύσεις με τη Βόρεια Κορέα για ένα συναφές θέμα όταν υποχωρεί και υπονομεύει τη συμφωνία με το Ιράν. Θεωρώ λοιπόν ότι η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών θα πρέπει να δείξει ότι έχει την ικανότητα, την βούληση να προχωρήσει ειλικρινά σε συζητήσεις ε, με τη Βόρεια Κορέα και ταυτόχρονα να έχει αντίθετη στάση με το Ιράν. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο σε δύο ακόμα συναδέλφους. Πολύ σύντομα παρακαλώ. Η Άννα Γκόμες και μετά ο κύριος Λίτς για να κλείσει προσωπώντας τον ε, εισηγητή. Ευχαριστώ. Όταν επισκέφθηκαν πρόσφατα το Ιράν, αντιπροσωπεία της Επιτροπής ΑΦΕΤ και της Υποεπιτροπής ΔΡΟΑ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μας ενημέρωσαν ότι γινόντουσαν διαδηλώσεις τότε, θυμάστε, ε, τέλη του 17, αρχές του 18 και μας είπαν ότι ε, ο λόγος ήταν η δυσφορία κατά της κυβέρνησης για την οικονομική διακυβέρνηση και για την ε, στρατιωτική περιπέτεια στην οποία έχει μπει το Ιράν στη Συρία. Και τότε μάθαμε λοιπόν ότι υπήρξαν σημαντικές επιπτώσεις και εσωτερικά για το καθεστώς από το γεγονός ότι οι Ισραηλινοί ε, βομβάρδισαν ε, σημαντικές Ιρανικές εγκαταστάσεις ε, στη Συρία και τις κατέστρεψαν. Σε ποιο βαθμό λοιπόν αυτό έχει επιπτώσεις στο ίδιο το Ιράν, στην εσωτερική πολιτική σκηνή και στις εξελίξεις Και πώς βλέπετε να διαχειρίζονται οι Ιρανοί αυτή ε, την αντίφαση. Έλεγαν οι ίδιοι ότι ήταν θύματα των χημικών που χρησιμοποιούσε ο Σαντάμ Χουσέιν στο Ιράκ και τώρα οι ίδιοι ενέχονται στην χρήση χημικών στη Συρία. Πώς μπορούν να το διαχειριστούν αυτή την εσωτερική αντίφαση. στο βαθμό που ακούγονται και κάποιες άλλες ε, φωνές και δεν υπάρχει μόνο καταστολή της ε, διαφωνίας και της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Λίτς. Ε- Σας ευχαριστώ. Όπως αναφέρατε τη διασκήψη ασφαλείας του Μονάχου και είπατε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι μόνο ο πρόεδρος. Θυμάμαι ότι κάποιος είχε πει, κύριος ότι άμα δει κανείς τα tweet ε, του κυρίου Προέδρου είναι σημαντικά, αλλά στη διάσκεψη ασφαλείας του Μονάχου συζητήθηκε και από τον Νετανιάχου αυτή η απειλή ε, αναφέρθηκε από το Ισραήλ ε, σε όλη την περιοχή, πόσο περίπλοκος είναι και ο ρόλος του Ιράν στην περιοχή, βλέπουμε. Το ζήτημα της Βόρειας Κορέας θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα Βλέπουμε πολλή κίνηση εκεί. Αν δείτε την επίσκεψη στην Κίνα, τις συναυλίες, ε, ε, τους Ολυμπιακούς, ε, συνεργασία Βορειάς και Νότιας Κορέας σε διάφορα θέματα. Ε, αυτό μας δείχνει ότι πρέπει να συνεχίσουμε ε, να παίξει σημαντικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση στο, Υπουργείο, στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών τη Δευτέρα. Τι θα γίνει θα μπορούσε να υπάρξει κάποιο άλλο σημείο, κάποια δήλωση που θα μπορούσε να αναφερθεί εκεί στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, κάτι για να δείξουμε ότι η Ευρώπη παίρνει σοβαρά αυτό το ζήτημα τη 12 η Μαου και ότι προβλέπουμε να αντιδράσουμε. Μια ερώτηση αναφερθήκατε στον τραπεζικό τομέα που είναι σημαντικό. Είχαμε και μια αντιπροσωπεία Ιρανών εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο που ήρθαν και τόνισαν ένα ζήτημα που είχε τονιστεί και στη διάσκεψη ασφαλείας του Μονάχου, τα περιβαλλοντικά ζητήματα στην περιοχή. Θα μπορούσε αυτό να υπάρξει ένα νέο κομμάτι των συνομιλιών. Αναφέρθηκε για το ζήτημα των αμοθιελών ε, στη διασκέψη ασφαλείας του Μονάχου από τους εκπροσώπους του Ιράν και είπαν ότι είναι διατεθειμένοι να κάνουν περαιτέρω συζητήσεις, συνομιλίες. Ε, να συζητήσουμε δηλαδή σε διπλωματικό επίπεδο τις αμοθύελε, τα ύδατα, διάφορα τέτοια ζητήματα περιβαλλοντικά που θα πρέπει να λάβουμε και αυτά υπόψη, διότι αισθανθήκαμε ότι είναι διατεθειμένα να τα συζητήσουν. Θα υπόσχομαι ότι θα είμαι σύντομη. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που είπατε για τους άλλους ε, παραγόντες στην Ασία, που θέλουν στενότερη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και περαιτέρω εξέλιξη των σχέσεων. Ε, εδώ στην αίθουσα, ξέρετε, έχουμε και το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας. Μην το ξεχνάμε, έχει ξεκινήσει κάτι. Ε, έχετε παρατηρήσει να υπάρχουν κάποιες εξελίξεις. Ευχαριστώ πολύ. Μόνο πέντε λεπτά θα σας δώσω το λόγο για να κλείσετε, παρακαλώ. Right, I will try. Mm, I don't actually need this now. Um, I will try. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Για την κοινή γνώμη στο Ιράν θα μιλήσω. Σε μια χώρα όπως το Ιράν είναι πολύ δύσκολο να αξιολογηθεί σωστά η κοινή γνώμη σε ολοκληρή τη χώρα. Ένα από τα βασικότερα πράγματα στο Ιράν είναι πόση επαφή πρόσβαση έχουν στα μέσα κοινωνική δικτύωση ε, οι άνθρωποι, ο λαό του Ιράν. Ε, κάποιοι άνθρωποι συνδέονται, γίνονται κάποιε συζητήσει, αλλά έχουμε περιορισμένη κατανόηση, θα πω επιφυλακτικά. Περιορισμένη εικόνα, αλλά οι ειδήσει που ακούμε και τα πράγματα που μαθαίνουμε για τις διαμαρτυρίες ε, στο Ιράν χαρακτηρίζονταν από κοινωνικο-οικονομικά θέματα και από πολιτική δυσαρέσκεια. Δυσαρέσκεια για τον πολιτικό κόσμο και κατά την άποψή μου παρατηρούμε ότι γίνεται μια συζήτηση δημοσίω στη χώρα που είναι κάτι καινούριο ε, για την τελευταία 30 ετία. ουσιαστικά. Ε, σχολιαστές, δημοσιογράφοι, καθηγητές πολλοί συζητούν διάφορα πράγματα. Πράγματα που ήταν ταμπού συζητώνται αυτή τη στιγμή. Ε, άνθρωποι οι οποίοι θεωρούνται βασικοί, σε βασικές εκλογικές περιφέρειες της Ισλαμικής Δημοκρατίας παρουσιάζουν νέα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και βλέπουμε στο επίκεντρο πολλές συζητήσεις για ε, οικονομικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα πρέπει να γίνουν άμεσα. Και όπως είπα νωρίτερα, αυτό αποτελεί τεράστιο πίεση ε, για τους κυβερνώντες. Θα πρέπει να λάβουν κάποιες δύσκολες αποφάσεις για το μέλλον, να δουν πώς θα καταμεριστεί η οικονομική και η πολιτική δύναμη και εξουσία στη χώρα. Σίγουρα υπάρχει και κάποια σχέση με τις διάφορες δράσεις του Ιράν σε χώρες όπως η Συρία, στο Λίβανο και αλλού. Και αυτό ήταν κομμάτι, το... ήταν θέμα στις διαμαρτυρίες και στα σλόγγαν που ακούστηκαν. Αλλά πιστεύω ότι το πιο δύσκολο, ε, αυτό που αναφέρθηκε περισσότερο από τους διαμαρτυρόμενους ήταν η... Ε, τα οικονομικά. Σχετίζεται με το ότι οι προσδοκίες ήταν πολύ υψηλέ. Περίμεναν ότι η συμφωνία για τα πυρηνικά θα είχε φέρει καλά αποτελέσματα, πράγμα το οποίο δεν συνέβη. Οπότε η κυβέρνηση θα πρέπει να αποκριθεί σε αυτό, θα πρέπει να δώσει και κάποια απάντηση. Όσον αφορά τις περιφερειακές συνομιλίες, την κλιματική διπλωματία, εγώ είμαι υπέρ τέτοιου είδου συνομιλιών. Ταξιδεύοντας και στην περιοχή πρόσφατα, μάλιστα πριν δύο εβδομάδες, έχω να πω ότι παρότι το Ιράν δηλώνει ότι είναι διατεθειμένο να κάνει τέτοιες συνομιλίες, άλλα μέρη τη συζήτηση στην περιοχή δεν είναι διατεθειμένα. Οπότε το Ιράν θα πρέπει να δημιουργήσει κάποια εμπιστοσύνη ώστε οι άλλοι περιφερειακοί του ΕΤΕΡΕ να δείξουν βούληση να συνεργαστούν. Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε απόψη ευρωπαϊκή είναι να πιέσουμε και να ενθαρρύνουμε όλες τις ε, πλευρές ε, για τη λήψη μέτρων ενθάρρυνσης της εμπιστοσύνης, παρότι δεν υπάρχει τέτοια όρεξη. Όρεξη υπάρχει για κλιμάκωση, για να το πω ειλικρινά. Κάτι πολύ ανησυχητικό. Και τέλος, όσον αφορά το ζήτημα της οικοδόμησης ε, ενός συνασπισμού, από όσο γνωρίζω δεν έχουν συμβεί και πολλά σε αυτό το μέτωπο. Εγώ το υπερασπίζω ως ιδέα. Ξέρω ότι γίνονται τακτικές συναντήσεις με συναδέλφους από την Ιαπωνία, την Νότιο Κορέα για το ζήτημα αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι έχουμε κάποια συλλογική δράση που θα οδηγήσει σε κάποια διαδικασία σχεδιασμού αντιμετώπισης εκτάτων περιστατικών. Θα κλείσω εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και πάλι, κύριο Σαντιμπάρ. Τρία πράγματα σύντομα. Αρχίζω από τη Βόρεια Κορέα. Και μετά θα πω δύο λόγια για το Ιράν, την εσωτερική κατάσταση και φυσικά την Ευρώπη. Για τη Βόρεια Κορέα. Όλοι σας, φαντάζομαι, όπως ε, και είπε και η ευρύτερη κοινότητα θεωρεί ότι το να αποχωρήσουν οι Ηνωμένε Πολιτείες από τη συμφωνία με το Ιράν λίγες μέρες πριν συναντήσουν τον Κιν Βιονκούμ δεν είναι καλό. Οι Αμερικανοί το βλέπουν διαφορετικά. Ακριβώς για να δείξουν πυγμή ε, στη ε, συζήτηση με το, τη Βόρεια Κορέα, καταγγέλνουν τη συμφωνία για το Ιράν, ε, θεωρώντας τη ασθενή, θεωρώντας ότι το Ιράν δεν την τηρεί ε, και τα λοιπά. Και το θεωρούν ακριβώς αυτό προαπαιτούμενο της έναρξης των συζητήσεων με τη Βόρεια Κορέα. Δεν λέω ότι συμφωνώ με την άποψη αυτή, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι επικρατεί μεταξύ των σκληρών πυρηνικών ε, στην Ουάσιγκτον για την εσωτερική κατάσταση στο Ιράν. Είναι πολύ έντονη συζήτηση, ε, ε, έτσι, παλόμενη η κοινωνία αυτή τη στιγμή ε, στο Ιράν. Οι Ευρωπαίοι βεβαίως θα πρέπει να ασχοληθούν με όλα αυτά τα θέματα, τα περιβαλλοντικά, τις κοινωνικές ανησυχίες, τις οικονομικές. Ήταν πολύ ψηλέ οι προσδοκίες, αλλά ακριβώς ο πύχης μπήκε τόσο ψηλά για να συμφωνήσουν οι διάφορες πλευρές ε, στο ε, Ιράν και ο ανώτατος ηγέτης ο ίδιος ε, και τώρα βλέπουμε ότι ήταν πολύ ψηλά ο πύχης και η απόδοση είναι μάλλον μικρή. Ακούστηκε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η ενθάρρυνση η οικονομική σε τομείς που δεν κυριαρχούνται από το δολάριο, δηλαδή και σε τίτλους που δεν εκδίδονται σε δολάρια. Τελικά όμως το Ιράν, η κοινωνία διψάει για περισσότερο άνοιγμα, για περισσότερη δικαιοσύνη και εσωτερικά στη διακυβέρνηση της χώρας. Και τέλος για την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης βεβαίως θα ήταν πολύ καλό εάν το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων τη Δευτέρα ε, κατέληγε κάπου δεν έχω εσωτερική πληροφόρηση, αλλά αν υπάρξει ένα ψήφισμα που λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται για το χειρότερο και λαμβάνει μέτρα αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων, αρκεί αυτό για τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για να δείξει στα άλλα μέρη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σοβαρή στάση και δέσμευση. Για το Brexit κάτι που ρώτησατε. Υπάρχει μια ε, λέξη δύσκολη να προφερθεί και ακόμα πιο δύσκολη να εφαρμοστεί ε, στα αγγλικά compartmentalization, δηλαδή αυτός ο κατακαιρματισμός. Ε, πώς κοιτάμε τους διάφορους τομείς χωριστά, ότι υπάρχουν κάποιοι τομείς στους οποίους έχουμε καταλήξει, έχουμε συμφωνήσει και εκεί η συμφωνία ε, τηρείται και κάποιοι άλλοι τομείς δεν έχουν συμφωνηθεί και είναι πιο δύσκολοι. Για το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 πλέον, εάν συμβεί αυτό και το Ηνωμένο Βασίλειο εκτός Ένωσης θα πρέπει ε, να ε, έχουν συνεργασία σε τομείς κοινού συμφέροντος όπως είναι η συμφωνία με το Ιράν. μπορούμε να δούμε τις συμφωνίες αυτές, όχι συνολικές, αλλά κατακαιρματισμένες στα κεφάλαια που συμφωνούμε να συνεργαζόμαστε στην περιφερειακή ασφάλεια, στα, ε, στην περιφερειακή ασφάλεια. Και όταν θεωρείται το Ιράν ε, ως παράγον ε, αποσταθεροποίηση στην περιοχή, ε, όπως υπάρχουν και πολλοί άλλοι, ε, θα το δούμε ξεχωριστά. Ε, πάντως αυτά τα καταλαβαίνουν κάποιες φορές και από περήφανοι λαοί και στην περιοχή. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο εμπειρογνώμονες. Ήταν πολύ σημαντική συζήτηση. Ευχαριστώ και τους βουλευτές. Ολοκληρώνεται εδώ η δημόσια κρόαση και το σημείο 3 και θα περάσουμε ε, αμέσως μετά. Και αλλάζει και η Προεδρία. Θα έρθει να προεδρεύσει τώρα ο κύριος Φρόιντ. Παρακαλώ. So good morning from my side. I'm taking... Καλημέρα σας και από πλευρά μου. Αναλαμβάνω εγώ να προεδρεύσω τώρα. Χαίρομαι που βλέπω τόσου πολλούς βουλευτές εδώ παρόντες. Μάλλον ο καιρός θα φταίει. Βλέπετε είναι χαρά Θεού έξω. Έχει ξεχυθεί ο κόσμος. Κανονικά θα σας έλεγα, λέτε λίγο πιο μπροστά όλοι, να μην είμαστε τόσο ε, αραιά. Αλλά από ό,τι φαίνεται στην Επιτροπή Άφετ δεν επιτρέπονται τέτοια πράγματα, οπότε ας το αφήσω καλύτερα. Σημείο 4. Συνολική και ενισχυμένη συμφωνία εταιρική σχέση μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομική Ενέργεια αφενό και των κρατών μελών του και τη Δημοκρατία τη Αρμενία αφετέρου. Η είναι ο κύριος Λάσλο Τόικερς και θα ήθελα να του δώσω αμέσω το λόγο. Θέλετε να μας πείτε κάποια πράγματα για τη συμφωνία αυτή. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, πριν σας παρουσιάσω το σχέδιο έκθεσής μου, θα ήθελα καταρχήν να εκφράσω την ικανοποίησή μου διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αρμενία έχουν προχωρήσει τόσο πολύ στις διμερείς τους σχέσεις, καθότι υπάρχουν βεβαίως ακόμη πολλές προκλήσεις. Θα ήθελα να χαιρετήσω την Αρμενία που γιορτάζει τα 2.800 χρόνια από την ίδρυση της πρωτεύουσας Ερεβάν, που είναι μια χριστιανική πόλη η οποία αντιστέκεται παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Γερμανία σήμερα, αντιμετωπίζει το παρελθόν του κομμουνιστικού της καθεστώσος, προκλήσεις δημογραφικές, δυσκολίες οικονομικές. Είναι όμως διατεθειμένη να βρει τρόπους να προχωρήσει, να γίνει μια ελεύθερη και σαφώς ευρωπαϊκή χώρα. Η συμφωνία αυτή, συνολική και ενισχυμένη, η οποία υπογράφει τον Νοέμβριο του 2017, μας ε, παρέχει ένα πλαίσιο συνεργασίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει προτεραιότητες σύναψη συμφωνιών με τις γειτονικέ χώρες, τις οποίες επικρατεί βεβαίως η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και ο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στα πλαίσια αυτά η σύσφυξη των σχέσεών μας με την Αρμενία σε μια δύσκολη και ταραγμένη περιοχή παραμένει ύψιστη προτεραιότητα. Στενή συνεργασία με την Αρμενία και με τις γειτονικές της χώρες που βασίζεται σε εμπιστοσύνη, σε διαφάνεια, παραμένει καθοριστικός στόχος για την ευημερία όλης της ε, περιοχής η γεωπολιτική μας και οι στρατηγικές μας επιλογές μας οδηγούν σε δέσμευση και στενές σχέσεις με τις γειτονικές μας χώρες. Εγώ λοιπόν σαν εισηγητής θα συνεχίσω τις προσπάθειές μου έτσι ώστε όλα αυτά να καθοδηγήσουν την δράση μας και τις προσπάθειές μας με έναν ουδέτερο και διαφανή τρόπο. Πιστεύω ότι ο συνάδελφος, ο κύριος Νικολάη, έχει και αυτός μια εξίσου εξισορροπημένη, συγγνώμη, ισορροπημένη προσέγγιση στις προσπάθειές του για το Αζερβαϊτζάν. Τώρα, όσον αφορά το κείμενο της έκθεσης αυτό καθεαυτό, υπάρχουν πολιτικές πτυχές και οικονομικές, τις οποίες θα σας παρουσιάσω. Καταρχήν, ο σεβασμός των θεμελιωδών αξιών, κράτος δικαίου, ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία, που αποτελούν, αν θέλετε, την καρδιά αυτής της ε, συμφωνίας. Θέλω η έκθεση αυτή να βασιστεί σε αυτές τις θεμελιώδες αξίες. Περαιτέρω πρόεδρος στις σχέσεις μας εξαρτάται καθοριστικά από το σεβασμό αυτών των θεμελιωδών αξιών. Οι εταίροι μας στην Αρμενία έχουν δείξει τη δέσμευσή τους και βεβαίως επιθυμούμε να συνεχίσουν να δεσμεύονται και να τηρούν αυτές τις θεμελιώδεις αξίες, όπως υπεγράφει στην Συμφωνία Πλαίσιο το Φεβρουάριο του 2018. Αυτά όλα αναγράφονται σε ένα ξεχωριστό παράρτημα της Συμφωνίας. Θα πρέπει να συνεχίσουν οι εσωτερικές μεταρρυθμίσεις, ιδιαίτερα η ομαλή μετάβαση από ένα προεδρικό σε ένα κοινοβουλευτικό σύστημα η κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να μπορεί να συνεχίζει να παίζει το ρόλο της στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Η κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να συνεχίσει να παρέχει συμβουλές και να συνεργάζεται με τη κυβέρνηση όσον αφορά το Ναγκόρνο Καραμπάχ και τους μετατοπιστέντες καθώς και την επιστροφή τους. Η έκθεση υπογραμμίζει την ανάγκη να συνεχίσει δέσμευση από μέρους των αρχών της Αρμενίας για να υπάρξει ειρηνική επίλυση αυτής της ε, διαφοράς. Στηρίζουμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση την ε, δράση της διεθνούς κοινότητας στα πλαίσια της ομάδας του Μίνσκ για την τήρηση αυτών των αρχών. Προτείνουμε κάποιες λύσεις οι οποίες να είναι κοινά αποδεκτές, αποδεκτές από τα δύο μέρη, έτσι ώστε να βρεθεί λύση κοινά αποδεκτή. Θεωρούμε ότι μια παρόμοια προσέγγιση θα πρέπει να επικρατήσει και στην έκθεση που αφορά το Αζερβαϊτζάν. Μια κοινά αποδεκτή επίλυση αυτής της διαφοράς σίγουρα χρειάζεται πολιτικό θάρρος και δέσμευση των ηγετών και της Αρμενίας αλλά και του Αζερβαϊτζάν. Δεύτερον, όσον αφορά την συνεργασία σε οικονομικό και εμπορικό επίπεδο, η έκθεση υπογραμμίζει την ευχή η ΣΥΠΑ να δώσει νέες ευκαιρίες και δυνατότητες στην Αρμενία, στους πολίτες της Αρμενίας, που ζουν στην Αρμενία ή που επιθυμούν να επιστρέψουν στην Αρμενία. Η έκθεση επίσης αναφέρεται στις δεσμεύσεις του ΠΟΕ αλλά και πέραν των δεσμεύσεων αυτών θέματα και τομείς όπως ε, τα πνευματικά δικαιώματα, η διαφάνεια, η πρόσβαση για τα ευρωπαϊκά προϊόντα, στις αγορές της Αρμενίας. Τώρα, όσον αφορά την ενέργεια, την προστασία του περιβάλλοντος, το Ερεβάν θα πρέπει να συνεχίσει την πρόοδο και την μείωση της εξάρτησης από την εισαγωγή ενέργειας καθώς και την ε, ανάπτυξη των δυνατοτήτων ε, της εσωτερικής αγοράς. Θα πρέπει εδώ να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μας στους τομείς αυτούς. Επαναλαμβάνω εξάλλου στην έκθεση τις ε, προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και την υποχρέωση να υποβάλουν οι αρχές της Αρμενίας κάθε εξάμεινο μια έκθεση πρόοδου για την υλοποίηση των δεσμεύσεων. Συνεχίζεται εξάλλου η διαδικασία παρακολούθησης. Όσον αφορά όλες σας τις προτάσεις, με μεγάλη χαρά θα τις εξετάσω και θα τις ενσωματώσω στην έκθεσή μου. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ, λέει και ο Πρόεδρος στα Ουγγρικά. Ε, επόμενος ομιλητής, ο κύριος Σόλτς, σκιώδης εισηγητής, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω ρητά τον εισηγητή για το έργο του και τον κόπο του ε, στο σχέδιο εργασίας και όλη τη διαδικασία εφαρμογής ε, ε, της συμφωνίας αυτής και διάνοιξη νέων διάβλων συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Αρμενίας. Θα ήθελα να τονίσω ότι ε, καταρχάς συμφωνούμε με τον εισηγητή στη βασική κατεύθυνση. Εγώ όμως θα κάνω και κάποιες τροπολογίες που αφορούν την ειδική θέση αυτής της συμφωνίας που θέλουμε να τονίσουμε. Δηλαδή η συμφωνία δεν θέτει ε, και να υπόψη μόνο το πλαίσιο, αλλά και την πολιτική, την πολυδιάστατη πολιτική, εξωτερική πολιτική της Αρμενίας και τη σεβόμαστε. Δηλαδή, συνεργάζεται με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και ε, στην Οικονομική Ένωση των Ουραλίων ε, συνεργάζεται, ε, που είναι πολύ σημαντικό αυτό για την ίδια την Αρμενία. Επίσης, θα κάνουμε τροπολογίες για το τι γίνεται με τη σύγκρουση εκεί στο ορεινό Καραμπάχ. Ε, και στον Αγκόρνο Καραμπάχ έχουμε αντίστοιχες απαιτήσει και από το Αζερβαϊτζάν. Θα πρέπει να ζητάμε τα ίδια και από την Αρμενία. Όπως ε, συζητήσαμε εδώ πριν από λίγες εβδομάδες ε, στην Επιτροπή μας με τον Υπουργό Εξωτερικών της ε, Δημοκρατίας της Αρμενίας. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να πιέσουμε ε, να δημιουργηθούν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, βιώσιμα και μόνιμα για να ξεπεραστεί αυτή η απροθυμία, η απόλυτη άρνηση συμβιβασμού, αυτό το, το τέλμα για να υπάρξει μια τελική οριστική συμφωνία ε, για κατάπαυση του πυρός, παρακολούθηση, ε, μη χρήση βίας, ε, αφοπλισμό των εμπλεκόμενων μερών κλπ. Και αμοιβαία θα πρέπει να δηλώσουν οι δύο πλευρές ότι δεν πρόκειται στο μέλλον να προβούν σε εχθροπραξίες για να υπάρξει οριστική ειρήνη για τα οικονομικά δυο λόγια, αν μου επιτρέπετε τώρα. Θεωρούμε απαραίτητο η Αρμενία να έχει μια ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη και να παραμείνει η προοπτική της και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και προς την άλλη πλευρά. Ε, και προς τη ρωσική ε, αγορά. Έχει συμφέρον η Αρμενία να είναι παρούσα. Υπάρχει Ευρωασιατική ε, Επιτροπή Οικονομικής Συνεργασίας και ποντάρει σε αυτή και ενδιαφέρεται η Αρμενία. Μας το έχουν πει και σε μας. Ένα θέμα που έχει να κάνει με το επόμενο, θα συζητήσουμε για τον ΟΗΕ, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η Αρμενία έχει υπογράψει μόνο ε, το καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και δεν το έχει κυρώσει. Ε, καλό θα ήταν να το κυρώσει όμως τώρα. Όπως συμφωνήθηκε ε, στην Καμπάλα στην Ογκάντα το 2010. Θα ήταν ένα παραπάνω βήμα ε, για ενίσχυση και σύσφυξη των διμερών ε, σχέσεων εξωτερικής πολιτικής και συνεργασίας. Ευχαριστώ και θα χαρώ για τη μελλοντική συνεργασία που θα έχουμε με τον εισηγητή και τους σκιώδες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σόλτς. Ο κύριος Στέτινα, επόμενος ομιλητής, παρακαλώ. Ευχαριστώ που δίνετε το λόγο κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον κύριο ε, Τέκες για την εκθεσή του. Εν συντομία, πιστεύω ότι στο συνοδευτικό ψήφισμα, σε αυτό το ψήφισμα, πρέπει να επιβεβαιώσουμε για άλλη μια φορά την ευρωπαϊκή υποστήριξη στους ε, συμπροέδρους της ομάδας ε, για την επίλυση ε, του, του, της σύγκρουσης διαφοράς των Αγγόνο Καραμπάχ βάσει των αρχών 2.0.0 ε, που περιλαμβάνουν μη ε, χρήση βίας, ε, αυτοκυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα. Όπως αναφέρεται και στο δικό μας ψήφισμα για την Ανατολική Γειτονία που υιοθετήθηκε το Νοεμβρίο του 2015. Ε, συγγνώμη, το 15, 15 Νοεμβρίου του 2017. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε κυρία Στέτινα. Η κυρία Κλαμούτη. Ευχαριστώ πολύ. Να προσθέσω τα σχόλια που ακούστηκαν. Πρώτα απ' όλα ότι καλωσορίζω τη συμφωνία και τους ισχυρότερους δεσμούς και την υποστήριξη που συνοδεύει τη συμφωνία αυτή. Επίσης, τώρα δεδομένου το σχολείο που ακούσαμε σε σχέση με τις νέες οικονομικές ευκαιρίες, που απορρέουν από την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας της ΕΠΑ και το ότι θα πρέπει να τις αξιοποιήσουμε στο έπακρο, να μην τις αφήσουμε στο χαρτί, αλλά να τους δώσουμε ζωή, να δράσουμε, να οικοδομήσουμε αυτούς τους δεσμούς, ε, τις σχέσεις με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ειδικότερα και με τη σύνδεση αυτών των πολύ ζωντανών οικονομιών. Επιπλέον, πιστεύω ότι η ΣΥΠΑ θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει την ενίσχυση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αυτές τις πτυχές της συμφωνίας. Συμφωνώ με τα σχόλια του εισηγητή. Πρέπει να διασφαλίσουμε ε, την επίτευξη αυτών των αποτελεσμάτων. Θα πρέπει επίσης εκεί να αποτυπώνται και τα δικαιώματα των, ε, των ανθρώπων, τα ατομικά δικαιώματα. Για παράδειγμα, προστασία της υγείας ε, και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας αν παρατηρήσει κανεί την ε, συμφωνία, θέλει να έχει ως δικαιούχου το σύνολο της κοινωνίας. Και αυτό με φέρνει στο τελευταίο μου σημείο που αφορά την επικοινωνία. Από άλλες συμφωνίες ε, έχουμε παρατηρήσει ότι είναι πολύ σημαντικό αυτή η συμφωνία να μην είναι απλά μια συμφωνία υψηλού επίπεδου μεταξύ κυβερνήσεως, ε, της αρμενικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι κάτι το οποίο θα κοινοποιηθεί, θα, ενημερω... θα, θα, αποτελέσει το αντικείμενο ενημέρωση προς το λαό της Αρμενίας, να γνωρίζει ο λαός της Αρμενίας το ότι υπάρχει, τι προσφέρει, ποια είναι τα ωφέλη και ποια είναι η εξέλιξη των ωφελών αυτών καθώς θα προχωράει η εφαρμογή αυτής της συμφωνίας. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια επικοινωνία ε, σε κάθε βήμα εφαρμογής αυτής της συμφωνίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κύριε Μούντι. Δεν ξέρω αν θέλει κανείς άλλο το λόγο. Δεν βλέπω. Α, κάτι ξέχασα, λέει κυρία Μούντι. Μιλούσα για την ασφάλεια και την υγιεινή, αλλά ε, φυσικά ε, ήθελα να πω και για την νομοθεσία για την ισότητα να ενταχθεί στην νομοθεσία της Αρμενίας ε, εσωτερική ενωμητάξη. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ προετοιμάζοντας αυτά ε, όλα, μπορεί να θυμάστε ότι είχε έρθει ο κύριος Έντουαρτ Ναμπαλτιάν, Ναμπαλτιάν Υπουργός Εξωτερικών ε, της Αρμενικής Δημοκρατίας, το Φεβρουάριο για τα Αλλαγή απόψεων. Και ορισμένοι από εσά μπορεί να θυμάστε ότι ασχοληθήκαμε κυρίως με περιφερειακά ζητήματα ε, και λιγότερο με την συμφωνία αυτή καθ' αυτή. Για να έχουμε συνέχεια και συνοχή στη θέση μας, θα ήθελα να πω ότι οι εργασίες μας ε, για την έκθεση αυτή γίνονται παράλληλα με μια άλλη εργασία της κυρίας Νικολάη για τις μελλοντικέ σχέσει και συμφωνία με το Αζερβαϊτζάν. Και για αυτά τα τρία κείμενα την ίδια μέρα θα γίνουν συνεδριάσει των σκιωδών και η συζήτηση. Θυμίζω, αύριο λίγη προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών στις 11 το πρωί, 13 Απριλίου, 11 η ώρα το πρωί. Ωραία. Και τώρα ερχόμαστε στη σύσταση προς το Συμβούλιο σχετικά με την 73η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Ε, τώρα είμαι σε κάπως δύσκολη θέση γιατί είναι δική μου η έκθεση και καλούμε να την παρουσιάσω από τη θέση του Προέδρου. Αυτό δεν προβλέπεται από το πρωτόκολλο και την ε, ε, εθιμοτυπία δεν είναι πάρα πολύ σωστό. Τι να κάνω, να, να καθίσω στην διπλανή θέση τώρα για να μην προεδρεύω. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Όπως κάθε χρόνο έχουμε αυτή την έκθεση που είναι μια ευκαιρία να παρουσιάσουμε τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και για τη σχέση μας με ε, τα Ηνωμένα Έθνη αλλά και για τα πιο πιεστικά και επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν τον ΟΗΕ. Πριν μπω όμως ε, στις λεπτομέρειες της εκθεσής μας, θα ήθελα σύντομα να αναφέρω ένα ζήτημα που δείχνει πόσο σημαντικά και πόσο περίπλοκα είναι τα ζητήματα. Μόλις προχθές το Συμβούλιο Ασφαλείας συζήτησε για αυτό που είναι μάλλον ε, επίθεση με χημικά όπλα στη Συρία και την αντίδραση του ΟΗΕ σε αυτές τις ε, ε, φερόμενες φρικαλαιότητες. Και όπως έχουμε ξαναδεί, μια υπερδύναμη έθεσε βέτο και μπλόκαρε το ψήφισμα. Κάθε πλευρά λοιπόν καταψήφισε τις προτάσεις της άλλης. Όταν ε, διαφωνούν οι ΗΠΑ με τη Ρωσία, υπάρχει πλήρης αδιέξοδο και ε, ο κόσμος ολόκληρο υποφέρει. Αυτό είναι ολέθριες συνέπειε του ΒΕΤΟ που είναι ένας μηχανισμός που χρειάζεται πηγόντως να αναθεωρηθεί και να μεταρρυθμιστεί. Βεβαίως εμείς υποστηρίζουμε ενεργά τον Γενικό Γραμματέα για να ε, μεταρρυθμιστεί το σύστημα των Αμένων Εθνών, να είναι πιο αποτελεσματικό για την ασφάλεια και την ειρήνη, πιο εστιασμένο και πιο επιχειρησιακό. Επίσης, υποστηρίζουμε το Γενικό Γραμματέα στις προσπάθειές του να κάνει ουσιαστικές αλλαγές έτσι ώστε το αναπτυξιακό σύστημα του ΟΗΕ να ευθυγραμμιστεί με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και τους στόχους ανάπτυξης για το 2030. Θέλουμε να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να αλλάξει η σύνθεση του Συμβούλου Ασφαλείας έτσι ώστε να αντανακλά καλύτερα το σημερινό κόσμο, ας πούμε να έχει μόνιμη έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας η Ευρωπαϊκή Ένωση. Φέτος Αποφύγαμε να ε, κατονομάσουμε την κάθε χώρα όπου σοβούν ε, διάφορες πολεμικές σειράξεις. Δεν το κάνουμε αυτό από συστολή. Αλλά ως μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών ε, ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα όλο το, το χρόνο. Και δυστυχώς οι ίδιες χώρες που αναφέρονται στην προηγούμενη σύνοδο, την 72η, δεν έχουν δει ειρήνευση στις συγκρούσεις τους. Και δεν τις επαναλαμβάνουμε. Σε ό,τι αφορά για τους πολέμους, δυστυχώς αυτό αφορά και άλλα πράγματα. Ας πούμε, τη σεξουαλική βία, το βιασμό που χρησιμοποιείται ακόμα ως όπλο και συνιστά έγκλημα πολέμου. Γι' αυτό ζητούμε πιο ενισχυμένη προστασία των γυναικών και κοριτσιών στις εμπόλεμες περιοχές. Σε ό,τι αφορά τα όπλα μαζικής καταστροφής και το θέμα της μη διάδοσης, υποστηρίζουμε όλες τις δράσεις του ΟΗΕ, ε, καθώς και ε, την πλήρη εφαρμογή ε, των συνδικών για τη μη διάδοση και καλούμε όλες τις χώρες μέλη του ΟΗΕ να υπογράψουν. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και να κυρώσω, για τα ανθρώπινα δικαιώματα βλέπουμε ότι περιστέλλεται η κοινωνία των πολιτών παντού σε πολλές χώρες στον κόσμο. Ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αδιέρετα, αλληλένδετα και αλληλοεξαρτώμετα. Να, όταν μιλούμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, στηρίζουμε το σύμφωνο για τους πρόσφυγες και για τους μετανάστες. Ε, θυμίζουμε έντονα στη διεθνή κοινότητα ότι χρειάζεται επαρκή χρηματοδότηση για την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ, έτσι ώστε να μπορεί να προστατεύει πλήρω και απολύτω πρόσφυγε ανά τον κόσμο. Και τελευταίο, χωρί αυτό είναι το λιγότερο σημαντικό, τονίζουμε και πάλι τη δέσμευσή μα προ το ε, σύμφωνα τη Συμφωνία για το Κλίμα του Παρισιού που θέλουμε να εφαρμοστεί παγκόσμια. Προβλέπω βλέπω και σε άλλες συστάσεις τη συνεδρία των συντονιστών, των σχεδόν μάλλον, και να σας θυμίσω ότι στις 25 Απριλίου στις 11 η ώρα λίγη προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχουμε διάφορους συναδέλφους που έχουν ζητήσει το λόγο. Ο κύριος Τόκες πρώτος. Εξ του κύριου Κοβάτσεφ. Ναι. Ο κύριος Κόβατσοφ μου ζήτησε να διαβάσω αυτό που έγραψε. Σαν εισηγητής των ε, δύο προηγούμενων εκθέσεων, τα Ηνωμένα Έθνη, θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Φρόιντ για την ε, σύνταξη αυτής της έκθεσης παρατηρούμε ότι εδώ δεν στοχεύεται ιδιαίτερα μια χώρα. Θα θέλαμε, αν μπορούσε ο εισηγητής να διασαφηνίσει ποιοι είναι οι στόχοι του για το τελικό κείμενο και αν θα υπάρξουν ε, όσον αφορά τις συγκεκριμένες χώρες τροπολογίες ή αν θα ενσωματωθούν οι αναφορές αυτές στο κείμενο της έκθεσης. Βεβαίως και υπάρχει ανάγκη για μία αναθεώρηση γενικότερη του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών καθώς και του Συμβουλίου Ασφαλείας και αυτό ενσωματώνεται στο πρώτο τμήμα της έκθεσης. Μία τέτοια μεταρρύθμιση σαφώς και θα πρέπει να οδηγήσει στην αναζωγόνηση του έργου και των δραστηριοτήτων της Γενικής Συνέλευσης καθώς και του συντονισμού της δράσης όλων των οργάνων των Ηνωμένων Εθνών. Όπως και στις προηγούμενες εκθέσεις, η ομάδα του ΕΛΚ θα ήθελε να επαναλάβει με σαφήνεια το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το θέμα του παγκόσμιου χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του αλληλένδετου χαρακτήρα αυτών και ότι ο σεβασμός αυτών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σαφώς θα πρέπει να στηριχθεί και να ενισχυθεί. Στα πλαίσια αυτά θεωρούμε ότι υπάρχει ένα κενό εδώ στο τμήμα που αναφέρεται στο κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και την ανεξιθρησκεία. Εμείς θα συνεχίσουμε να συνηγορούμε υπέρ της ανεξιθρησκείας. Επίσης θεωρούμε ότι ένα σημαντικό τμήμα της έκθεσης που είναι η καταπολέμηση της ε, τρομοκρατίας λείπει από την ε, ετήσια έκθεση, κάτι που σίγουρα θα πρέπει να ενσωματωθεί. Θεωρούμε ότι είναι καθοριστική σημασίας. Για την ομάδα του ΕΛΚ θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να επαναλάβουμε για άλλη μια φορά την ε, καταδίκη κάθε τρομοκρατικής δράσης. Η εξάλληψη των τρομοκρατικών οργανώσεων είναι απαραίτητη, ιδιαίτερα όσον αφορά το ISIS και το Daesh. το θέμα του ορισμού των κλιματικών προσφύγων και τη συζήτηση περί αυτό τον ορισμό. Η ομάδα του ΕΛΚ δεν θα ήθελε να ανοίξει η συζήτηση αυτή, καθότι είναι μια συζήτηση δύσκολη για την ομάδα του ΕΛΚ. Για τα θέματα της συνευτικής διαδικασίας αναφέρεται κάπου η Αφρικανική Λίγα. Βλέπουμε όμως ότι δεν αναφέρονται άλλοι διεθνείς οργανισμοί. Ολοκληρώνω το σχέδιο έκθεση αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή βάση για περαιτέρω συζήτηση και συμβιβασμό και για την ψηφοφορία στην Ολομέλεια αργότερα μέσα στο 2018. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριε Τόκερς. Θα επανέλθω στα σημεία που αναφέρατε και θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Σόλτς που είναι σκιώδης. Όχι. Όχι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μου δίνετε το λόγο πρώτα και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω για την uh, συστάση αυτής της έκθεσης. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και προκλητικό το θέμα. Συμφωνώ μαζί σας ότι βρισκόμαστε σε μια καθοριστική στιγμή και προσπαθούμε να συντάξουμε τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν την ε, Γενική Συνέλευση που θα πρέπει να λάβει υπόψη της όλες αυτές τις διεθνείς προκλήσεις που δυστυχώς χαρακτηρίζονται από σημαντικές απειλές όχι μόνο σε περιφερειακό επίπεδο αλλά και παγκοσμίως. Γι' αυτό και εγώ θα πρότεινα να υπάρξει σύνδεση αυτών των προκλήσεων με τις σημαντικές αποστολές και στόχους των Ηνωμένων Εθνών που έχουν σαν σκοπό να ενσωματωθούν αυτές τις προκλήσεις και στην ε, ατζέντα για βιώσιμη ανάπτυξη και βεβαίως την υλοποίηση των 18 στόχων που εμπεριέχονται σε αυτή την ατζέντα. Με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά περιγράφουμε με ακρίβεια με ποιο τρόπο μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και οφείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεισφέρει με δραστήριο τρόπο, με ενεργητικό τρόπο σε αυτήν την υλοποίηση. Και αυτό για θέματα ασφάλειας, για τις ειρηνευτικές διαδικασίες, πρόληψη των συγκρούσεων, και βεβαίως την ενεργοποίηση των ε, εργαλείων και μέσων που διαθέτουν τα Ηνωμένα Έθνη. Περισσότερη δράση για θέματα διάθεσης των εξοπλισμών, αντιμετώπισης όλων των στόχων που αφορούν τους πρόσφυγες, ε, τους ε, μετανάστες. και διάφορες άλλες δραστηριότητες που πρέπει και μπορεί να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα του κλίματος, της ε, διπλωματίας γύρω από το κλίμα και βεβαίως τμήματα αυτής της έκθεσης θα πρέπει να επεξεργάζονται και θέματα ανάπτυξης, οικονομικά θέματα. Και ενίσχυση της ε, διεθνούς οικονομικής συνεργασίας με ένα πιο υπεύθυνο και σωστό τρόπο. Θα θέλαμε λοιπόν να συνεχίσουμε σε στενή συνεργασία με εσά, κύριε Σιγητά, την επεξεργασία του κειμένου αυτού και ελπίζουμε να έχουμε περαιτέρω δυνατότητες συνεργασίας μαζί σας, εμπλουτισμού του κειμένου. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σόλτς, κυρία Λόπη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, και ε, Ευχαριστώ κύριε εισηγητή. Είναι πολύ καλή έκθεση θεωρούμε. Επισημαίνει τα σημαντικότερα θέματα στα οποία θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην επόμενη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης. Όσον αφορά τις δικές μας τροπολογίες, θα κάνουμε αναφορά στην απειλή ε, που προέρχεται από την πολυμερή αντιμετώπιση και θα εκφράσουμε την άποψή μας για τα πολυμερή συστήματα. Θέλουμε επίσης να υπογραμμίσουμε το πόσο σημαντικό είναι να μιλά σε τέτοια φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση με μία φωνή. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έλλειψη ενότητα μεταξύ των κρατών μελών, η οποία αποδυναμώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Ηνωμένα Έθνη. Επίση, θα υποβάλουμε τροπολογίε για περισσότερη έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα, τον τρίτο πυλώνα του χάρτη των ανθρώπινων δικαιωμάτων, που είναι και προϋπόθεση. Το Συμβουλίο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Δανίας είπε ότι πολλοί από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης βασίζονται στην πρόοδο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κάτι που θα πρέπει να θέσουμε λοιπόν στο επίκεντρο των Ηνωμένων Εθνών. Επίσης θα προτείνουμε να προσθεθεί ένα ε, δευτερεύον τμήμα για την βιώσιμη ανάπτυξη. Επειδή είναι ένας ε, τομέας ε, τον οποίο αμφισβητούν ορισμένα κράτη-μέλη ορισμένες κυβερνήσεις. Όπως είπε και ο κ. Σόλτσο, πρέπει οπωσδήποτε να υπογραμμίσουμε τη δέσμευσή μας να επιτύχουμε ε, τους στόχους αυτού του θεματολογίου του 2030. Θα υποβάλουμε και μια τροπολογία που θα σχετίζεται με το θεματολόγιο ειρήνης, τη νέα πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των να συμπεριλάβει τις φωνές των νέων στην πρόληψη ε, και στην οικοδόμηση της ειρήνης. Επίση, θα υποβάλουμε μια τροπολογία για την πρωτοβούλια περιβαλλοντικών δικαιωμάτων, την οποία καλωσορίζουμε αυτή την πρωτοβουλία των ΗΕ και ελπίζουμε να την υποστηρίξετε. Τέλος, για το Συμβουλίο Ασφαλεία των ΗΕ θα κάνουμε επίσης αναφορά σε διάφορες περιοχές όπου έχει να παίξει κάποιο ρόλο ο Οργανισμό των Εθνών ως ειρηνευτικός Αυτά προσβλέπουμε στην περαιτέρω συνεργασία μας. Θεωρούμε ότι θα είναι πολύ καλή έκθεση. Ευχαριστούμε. Κυρία Μούντι, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Αυτό που περίμενα ακριβώς από εσά, εξαιρετική, εξαιρετικό έκθεση. έκθεσης. Ένα-δυο σημεία τη εκθέση να αναφέρω. Πρώτα απ' όλα το Συμβούλιο Ασφαλεία των ΗΠΑ. Το είπατε στα εναρκτήρια σχολεία σα. Ναι, χρειάζεται μεταρρύθμιση ώστε το Συμβούλιο Ασφαλείας να είναι πιο αποτελεσματικό σε σχέση με τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε παγκοσμίω αυτή τη στιγμή. Δεύτερον, χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτή την προτεραιότητα που δίνεται στο ρόλο των γυναικών μέσα στην εκθεσή σας για την πρόληψη των ε, σειράξεων και για την αποκατάσταση μετά από σειράξεις. Εγώ θα υποβάλω τροπολογίες ε, που θα σχετίζονται με την άμεση συμμετοχή των γυναικών σε ειρηνευτικές διαδικασίες. Από τα ελάχιστα στοιχεία που έχουμε είναι απόλυτα σαφές ε, πόσο μακροχρόνια αποτελέσματα και βιωσιμότητα χαρακτηρίζει τις ειρηνευτικές διαδικασίες όπου έχουν συμμετάσχει γυναίκες. Όσον αφορά το κομμάτι της μη διάδοσης και τις σχετικές παραγράφους, δεδομένων των τελευταίων εξελίξεων ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο και τελευταία στη Συρία και πιο συγκεκριμένα τη χρήση των χημικών όπλων, Χαίρομαι που έχει συμπεριληφθεί αυτή η αναφορά. Τώρα, και από την προηγούμενη συζήτηση κατά πόσο αξίζει να συμπεριλάβουμε κάποια αναφορά στην JCPOA. Αυτό αναρωτιέμαι. Να τη συμπεριλάβουμε στην έκθεση. Και τέλος, ήθελα να συμφωνήσω και εγώ με την υποστήριξη που εξέφρασαν και οι υπόλοιποι για το τελευταίο σας σημείο το... Ε, την έκκληση αυτή για να γίνει κάποια συζήτηση για τους κλιματικούς πρόσφυγες, να υπάρξει ένας νομικός ορισμός στο μέλλον. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε και να επιδιώξουμε ε, περαιτέρω εξέταση αυτού του σημείου και να το αναφέρουμε και στην έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και ο Πρόεδρος τώρα ε, θα ζητήσει από τον εισηγητή να πει δύο λόγια. Είναι ευγνώμων για όλα τα συγχαρητήρια και τους επένους που άκουσα από εσά παρότι χάσατε κάποια θέματα που αναφέρονται στην έκθεση, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα φαντάζομαι κάτι που θα γνωρίζετε περισσότεροι. Ε, έχουμε περιορισμένο χώρο. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να προσέχουμε. Αν είχατε δει την αρχική έκθεση, ήταν τριπλάσια σε μέγεθος και περιλάμβανε τις περισσότερες από τις επιφυλάξεις που εξετάσετε, τις χώρες που αναφέρατε, το πρόβλημα με τις χώρες είναι ότι αν αναφέρει κανείς 4 ή 5, μετά κάποιος άλλος λέει γιατί αναφέρετε την, ε, την 6 και την 7 και όχι τις άλλες. Ε, έχουμε περιορισμού χώρου. Γι' αυτό παραλείψαμε κάποιε χώρε. Αλλά επίση ξέρουμε ότι και εσεί στι τροπολογίε έχετε το δικαίωμα να πάρετε τι χώρε που θέλετε και να αναφέρετε τι χώρε που θέλετε να συμπεριλαμβάνετε στην τελική έκθεση. Αυτό αφορά φυσικά και την καταπολέμηση τη τρομοκρατία. που παραλείψαμε φέτος παρότι υπάρχει σε κάθε έκθεση. γιατί έπρεπε να συμπεριλάβουμε κάτι άλλο. Αυτό που είπε την κυρία Μούντι, το τη συμμετοχή των γυναικών, τη σημαντική συμμετοχή των γυναικών στις ειρηνευτικές διαδικασίες. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και έχουμε ξανακάνει αυτή τη συζήτηση. Και ε, προηγήθηκε και η συζήτηση της, ε, για την JCPOA ε, σε σχέση με την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν οι γυναίκες έχουν διαδραματίσει ε, σημαντικότατο ρόλο ε, στη σύνταξη αυτής της συμφωνίας, όπως γνωρίζουμε όλοι, τόσο από ευρωπαϊκής όσο και από Ιρανική πλευράς και διεθνώς. Χαίρομαι λοιπόν ε, που είπατε ότι θα συμπεριλάβετε κάποια σχόλια, κάποιες παρατηρήσεις για αυτό το ζήτημα, κάποια ισχυρότερη διατύπωση. Ευχαριστώ για τη ζωηρή συζήτηση που κάναμε εδώ. Και να σας υπενθυμίσω ότι η προθεσμία για την υποβο... κατάθεση τροπολογιών είναι 25 Απριλίου. Έχουμε τώρα. Uh, next uh, is then in camera. Α, έχουμε και κλεισμένο το θηρόν συνεδρίαση. Θα αλλάξει τίποτα <laughs> ως προς τη συμμετοχή. Για να δούμε. Μπορεί. Uh, for all members of the European Parliament to be present. Παρακαλώ να παραμείνουν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όσοι δικαιούνται και οι υπόλοιποι να αποχωρήσουν.